Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε χθε. Και θα περάσουμε στην παρουσίαση της έκθεσης ε, της αποστολής μας στις Αζόρες που έγινε 2 με 5 Νοεμβρίου. κυρία Ριμπέρο, η κυρία Σοφία Ριμπέρο είχε οργανώσει αυτή την αποστολή της Επιτροπής Άγκρη στις Αζόρες ε, σε συνεργασία με τον κύριο Ρικάρντο Σάντος. Είχαμε χάρη στην αποστολή αυτή μια εξαιρετική ευκαιρία να διαπιστώσουμε η διεισόμαση τις ιδιαιτερότητες της ε, γεωργίας της Αζόρες και την ε, μεγάλη της εξάρτηση από τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στην περιοχή αυτή ε, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά η κτηνοτροφία και η γαλακτοπαραγωγή. Μέλη της αντιπροσωπείας ήταν ο κύριος Αντρία, ο κύριος Βοητσεχόφσκι, ο κύριος Αλμπερντές, Γιάννης Κίσεκε και Μιγγέλ Βιέγκας. και οι Θα ακούσουμε τώρα την ενημέρωση από την αποστολή αυτή, γιατί η έκθεση σας έχει ήδη μοιραστεί. Η κυρία Ριμπέρο θα μας κάνει μια, ένα σύντομο απολογισμό αυτής της αποστολής της Αζόρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας εκφράσω την τεράστια ικανοποίηση και την περηφάνεια μου για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τα πορίσματα της αντιπροσωπείας μας στις Αζόρες. Εκεί διαπιστώσαμε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η παραγωγή γάλακτος στην περιοχή αυτή. Και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν μέρος στην αντιπροσωπεία. Να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο Σεκέρσκι και τον Αλμπερντές, τον συντονιστή του ΕΛΚ, για την προσπάθεια που έκανε για να γίνει πραγματικότητα η αποστολή αυτή. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τους βοηθούς μου, τον Χέραλτ ε, του ΕΛΚ και τον Κοσάλβο και όσους συνέβαλαν σε αυτή την ε, αντιπροσωπεία. Φαίνεται από την έκθεση τεράστιες δυσκολίες που έχουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, για την γεωρική τους δραστηριότητα και παραγωγή. Ιδιαίτερα στις Αζόρες οι κλιματικές, μετεωρολογικές και γεωγραφικές στις συνθήκες δημιουργούν πολλές ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Βέβαια ε, έχουν, καταλήγουν και μια, σε μια παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας. Μάλιστα με το ρωσικό εμπάργο φάνηκε η τροτότητα αυτής της τοπικής οικονομίας που εξαρτάται κυρίως από τη γαλακτοπαραγωγή. Βέβαια το θέμα και το πρόβλημα δεν είναι αμυγός οικονομικό. Είναι και οικογενειακό και κοινωνικό γιατί αφορά την απασχόληση στις εξόχω απόκεντρε και περιφερειακές περιοχέ, αφορά τη βιοπικιλότητα, το σεβασμό του περιβάλλοντος, τη δυνατότητα αντοχής και επιβίωση της γεωργίας για ιστορικούς και πολιτιστικούς ε, λόγους. Είδατε ότι στις φλέβες ε, των κατοίκων των Σαζόρας ε, ρέει γάλα. Ε, είναι τεράστια εξάρτηση από τον κλάδο αυτό και θα ήταν κρίμα να χαθεί αυτή η μακροχρόνια παράδοση. Χρειάζεται να αντιδράσουμε για να επιβιώσει αυτή η παραγωγή, γιατί οι συνθήκες είναι αντίξωες και η καιρή χαλεπή για όλους. Ε, μερικοί θα καταφέρουν να ξεφύγουν από την κρίση, για άλλους όμως δεν θα είναι τόσο εύκολο όπως για τους παραγωγούς της Αζόρες βέβαια από μια θετική διάκριση μερικοί θα βγουν χαμένοι. Δεν ζητούμε αυτό. Θέλουμε απλώς να τηρηθούν οι συνθήκες και κυρίως το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει έκτακτα μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή με όλους τους περιορισμούς που έχουμε, δεν έχουμε καταφέρει ε, να έχουμε παραγωγή με ίσες ε, συνθήκες με τις υπόλοιπες περιφέρειες και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Φαίνεται από την έκθεση το τεράστιο κόστος μεταφοράς και για, τη, για, τα, την πρώτη ύλη και για τα μεταποιημένα προϊόντα. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης του κλάδου. Ζητώ όμως και τη δική σας υποστήριξη για να βελτιωθεί η εφαρμογή του ειδικού προγράμματος ε, της Γεωργίας ε, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το ΠΟΣΕΙ, που θα αναθεωρηθεί το 2017. Και τέλος, θα ήθελα να σας δώσω ένα μικρό δείγμα του πολύ ποιοτικού γάλακτος των Αζωρών. Ε, παραγωγής Unilate, ενός τοπικού γεωργικού συνεταιρισμού. Ελπίζω να το απολαύσετε. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σάντος και για ένα διαδικαστικό πρώτο στον κύριο Σελιμόβιτς. Πρώτα στον κύριο Σελιμόβιτς για το διαδικαστικό και μετά στον κύριο Σάντος. Ευχαριστώ. Θέλω να θέσω ένα θέμα που έχει θυγεί και πριν, το ξέρω. Ανησυχώ όμως που οι συνεδριάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επιτροπής Γεωργίας διεξάγονται ταυτόχρονα. Δημιουργεί πρόβλημα για μας που Είμαστε μέλη και των δύο επιτροπών, δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα και στις δύο. Αλλά δημιουργείται και πρόβλημα για μας που παρακολουθούμε τα θέματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και που επηρεάζονται και από αυτά που συζητούμε εδώ. Σήμερα συζητούν την έκθεση για την ΕΦΤΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και για μας αυτή την Επιτροπή. Ξέρω ότι το θέμα είχε τεθεί επιτάπητος Υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα ήθελα να θέσω την ιδέα, αν την στηρίζουν και άλλοι. Ας μην έχουμε όλες τις συνεδριάσεις σε διαφορετικές ώρες, αλλά κάποιε από αυτές που αφορούν ε, θέματα που είναι σημαντικά για μα και τα συζητούν και στι δύο επιτροπέ. Ο κύριος Σάντος τώρα γιατί ο κύριος Σελίμοβιτς έθεσε ένα διαδικαστικό οργανωτικό θέμα. Ο κύριος Σάντος για την αποστολή στην Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, κατάλαβα ότι ήταν διαδικαστικό το θέμα του κυρίου Σελίμοβιτς. Θα ήθελα και εγώ να διατρανώσω τη σημασία που είχε η πραγματοποίηση αυτή τη επίσκεψη της Αζόρες για το γεωργικό τομέα και το τομέα παραγωγής και να ευχαριστήσω θερμά τους βουλευτές και τους βοηθούς που συμμετείχαν στην εύρυθμη οργάνωση αυτής της αποστολής. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Μάκη Κόλταρ που από την ΕΣΥΝΤΕ μας βοήθησε στη διαδικασία αυτή και τους βοηθούς μου και τους συνεργάτες μου και κυρίω την Άννα Καμίλα που συνέβαλε τα μάλα στην διοργάνωση της επίσκεψης της αντιπροσωπείας και να ευχαριστήσω και τον βουλευτή Νονοτομέα από τις Αζόρες. Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να δούμε τα μάτια τους στην πραγματικότητα της γεωργίας των Αζωρών, που είναι πολύ διαφορετική και ιδιαίτερη σε σχέση με την υπόλοιπη υπηρετική γεωργία κατά κάποιο τρόπο. Φυσικά η αντιπροσωπεία μας επικεντρώθηκε στο γαλακτοκομικό τομέα που είναι ο πιο σημαντικός τομέα στην γεωργία των Αζωρών και έχει μεγάλη οικονομική σημασία. Ο κλάδος όμως αυτός, ο γαλακτοκομικός, έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα και από το ρωσικό εμπάργο που δημιουργεί προβλήματα στη γαλακτοπαραγωγή στην Ευρώπη και επίσης ε, με την εκπνοή των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων που επίσης επηρέασε την ε, παραγωγή γάλακτος παντού αλλά και στις αζόρες ιδιαίτερως. Έτσι αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από αυτούς τους δύο επιβαρυντικούς παράγοντες η παραγωγή μας. Επίσης, εξαιτία ε, των γεωγραφικών συνθήκων, της απομάκρυσης και του νησιωτικού χαρακτήρα αυτής της περιφέρειας, το κόστος παραγωγής είναι πιο υψηλό. Είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή γάλακτος στις Αζόρες από ότι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της υπηρετικής Ευρώπης. Γι' αυτό και ήταν απαραίτητα κονδύλια που δόθηκαν ε, στους παραγωγούς. Και μάλιστα αυτά τα κονδύλια φορούσαν κανονικές συνθήκες. Εδώ όμως δεν έχουμε πια κανονικές συνθήκες. Έχουμε συνθήκες κρίσης που μαστίζει ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει έτσι να αποθαρρυνθεί η τοπική οικονομία και κυρίως η παραγωγή γάλακτος παρά τις κρίσιμες συνθήκες. Και ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει η ευημερία των ζώων, η διασφάλιση των βοσκοτόπων και η υγεία και προστασία των ζώων. Η σημασία του γαλακτοκομικού κλάδου στις Αζόρες συνέβαλε στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και στην παραμονή του πληθυσμού στην Ήπεθρο και κυρίως ε, και νέων γενιών. Γιατί πρόκειται για ένα τομέα που στις Αζόρες ε, ε, έχει μέσω ηλικίας 10 χρόνια μικρότερο από ό,τι στην υπηρετική Ευρώπη. Βέβαια, όπως σας είπα, οι δυσκολίες είναι πολλές. Γιατί επειδή γίνεται επιλογή υπέρ της διαφοροποίησης, μειώνεται η ωφέλιμη γη σε υψηλά ε, σε, σε υψόμετρα άνω των 250 μέτρων. Είναι ορεινέ όμω οι περιοχέ των Αζωρών και μάλιστα θεστιογενεί. Οπότε οι γεωργικές συνθήκες είναι πολύ διάζωσε. Αυτό που φάνηκε από την επίσκεψη είναι ότι οι ιδιαιτερότητε των Αζωρών δικαιολογούν διαφοροποιημένη μεταχείριση. Επίσης ε, φάνηκε πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ και τα διαρθρωτικά ταμεία για την ανάπτυξη του κλάδου. Ο γαλακτοκομικός κλάδος είναι σήμερα πιο εύρωστος χάρη στα ταμεία αυτά. Μέχρι στιγμής έχει αντέξει στα πλήγματα. Αν και πολλοί παραγωγοί δυστυχώς έχουν εγκαταλείψει ε, την παραγωγή τους, παρόλο που όπως σας είπα το μέσα αυτός απασχολεί πολύ κόσμο και κυρίως νέους κτηνοτρόφους και παραγωγούς. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διαφυλαχθεί αυτός ο γεωργικός ιστός σε μια περιοχή που εκτός από την γαλακτοπαραγωγή έχει και σημαντικό τουρισμό και έχει σημειώσει αρκετή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντριέ και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Σεκέσκη, για την προσήλωση την οποία έδειξαν στο θέμα αυτό και τον ενθουσιασμό τους στη συμμετοχή της ε, αποστολής. Ελπίζω μετά την επίσκεψη αυτή να διαμορφώσετε καλύτερη γνώμη για την πραγματικότητα που επικρατεί στις και την ανάγκη ε, στήριξης των παραγωγών της. Αυτά και ελπίζω η επίσκεψη να αποτελέσει καλή βάση και για τις μελλοντικές μας εργασίες. Και μάλιστα η έκθεση για το γάλα που, του κυρίου Νίκολσον που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει ειδική μνήμα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδιαίτερα στην περιοχή των Αζωρών. Έχουμε καθήκον ως ευρωβουλευτές και κυρίως μέλη της Επιτροπής Άγκρη να επισημάνουμε τη σημασία αυτού του κλάδου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, δύο συνάδελφοι μας ζήτησαν το λόγο που έλαβαν μέρος και στην αντιπροσωπεία. Ο κύριος Αντρία και ο κύριος Δέσ. Ο κύριος Αντρία πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε η κυρία Ριμπέιρο και ο κύριος Σάντος. Η ποιότητα της επίσκεψης ήταν ε, υψηλή και ευχαριστώ και τους δύο και την ομάδα τους για τη διοργάνωση της επίσκεψης. Η επίσκεψη μας επέτρεψε να κατανοήσουμε τι σήμαινε ο ορισμός που χρησιμοποιούν στα ζώρες της ευτυχούς αγελάδας. Δηλαδή είδαμε τις εκμεταλλεύσεις είδαμε και πώς ε, συμβάλλει την κτηνοτροφία στα οικονομικά. Είδαμε τι σήμαινε αυτή η έννοια και θα ήταν σημαντικό να επιτρέψουμε στον κύριο Χόγκαν, τον επίτροπό μας, να πάει να δει, να καταλάβει τι είναι αυτού του είδους εκμεταλλεύσεις και τι αντίκτυπο ε, έχει η κρίση του γάλακτος. Όταν απευθυνόμεθα στους γεωργούς βλέπουμε ότι έχει αντίκτυπο μεγάλη ε, κρίση στην τοπική οικονομία. Η ποιότητα των γεωργών και των εκπροσώπων που συναντήσαμε καταδεικνύει πόσο είναι σημαντικό να αναδιοργανωθεί ο τομέας για να διατηρηθεί, να διαφυλαχθεί η τοπική οικονομία. Το, το είδαμε σε αυτή την υπερπεριφερειακή περιοχή πόσο σημαντική είναι η ιδιαιτερότητα. Στα εννιά νησιά του αρχιπελάγους είδαμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την αγορά και την παραγωγή βασικέ δυσκολίε και όσον αφορά την κινητικότητα. Έχουμε ευθύνη για αυτές τις υπερπεριφερειακές ζώνες και εκεί υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Οι δυσκολίες δημιουργούν προβλήματα για, όσον αφορά την κινητικότητα τις μεταφορές στο αρχιπέλαγος και πώς διασυνδέεται με την υπηρετική Ευρώπη το αρχιπέλαγος. Δημιουργούνται προβλήματα. Αυτά που είπε η κυρία Ριμπέρο και ο κύριος Σάντος δείχνουν ότι πρέπει να δούμε τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται τα προγράμματα και να προσαρμοστούν αυτά τα προγράμματα σε αυτού του είδους τις περιοχές. Ε, το πως θα εξεταστεί την επόμενη χρονιά η επίσκεψη μας επέτρεψε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προγράμματα. Αυτό το αρχιπέλαγος είναι ιδιαίτερο, έχει ιδιαιτερότητες και για την πολιτική της Ένωσης και γενικά για τη συγκεκριμένη περιοχή και γενικά για την προσέγγιση που ακολουθούμε για τις απόμακρες υπερπεριφερειακές ζώνες. Έχουν πολλές ιδιαιτερότητες οι Αζόρες. Αυτό ανακαλύψαμε στην επίσκεψη. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Αλμπερντές τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την Σοφία Ριβέιρο καθώς και τον κύριο Σάντος και τους συνεργάτες τους για την ε, καλή διοργάνωση του ταξιδιού. Εμείς στη Γερμανία λέμε ότι με τα ταξίδια μορφώνεται κανείς και πράγματι το ταξίδι αυτό συνέβαλε στην μόρφωσή μου πολλές ώρες από τη Λισαβόνα μέχρι, τους, ε, μέχρι τις Αζόρες και βλέπουμε με τον τρόπο αυτό, είδαμε δηλαδή με τον τρόπο αυτό πόσο μακριά είναι από την υπηρετική Πορτογαλία και αντιλαμβάνομαι έτσι και τον προβληματισμό που, ε, ή τα προβλήματα των νησιών αυτών. Δηλαδή προκύπτει και υψηλό κόστος για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Κάτι που ήταν σημαντικό για μένα είναι ότι τα νησιά αυτά αποτελούν μόνο το 2% της συνολικής έκτασης της Πορτογαλίας, παρόλα αυτά παράγουν το 30% το, της παραγωγής γάλακτος. Βλέπει κανείς δηλαδή πόσο σημαντική είναι η κτηνοτροφία και η γαλακτοπαραγωγή. Εάν δηλαδή πρόκειται τώρα να καταργηθούν προγράμματα, ίσως χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες ενισχύσεις λόγω της μεγάλης απόστασης από τον κορμό της χώρας. Κάτι άλλο που με εντυπωσίασε ήταν και πολύ υψηλές τιμές των ε, εδαφών. 75.000 ευρώ ανά εκτάριο. Δηλαδή αυτό σημαίνει πολύ υψηλές ε, τιμές και πολύ ψηλό κόστος και για την παραγωγή. Άλλο είναι και ο κατακαιρματισμός των εδαφών, διότι συχνά τα εδάφια που ε, βόσκουν οι αγελάδες είναι μακριά από τις εκμεταλλεύσεις. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, όντω καθώς και την μακρά απόσταση από την Μητροπολιτική Πορτογαλία και από τον ε, υπηρετικό κορμό της Ευρώπης, για να μπορέσουν οι εκμεταλλεύσει αυτές να παραμείνουν αποδοτικέ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τι άλλε και τους άλλους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ε, αποστολή που για μένα ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ε, δεν ξέρω, είχαμε πει πρόβλημα με τη διερμηνία, δεν ακουγόταν όλες οι καμπίνες. Εντάξει τώρα. Tak? dziękuję Σας ευχαριστούμε κύριε Ντές. Θέλει κανείς το λόγο παρακαλώ. Wenn der Kopfhörer nicht funktioniert hat, möchte ich nochmal wiederholen, dass ich mich bei unserem Εάν δεν λειτουργήσε η ε, διερμηνία, το μόνο που θέλω να πω, που λειτουργήσε βεβαίω, είναι ότι ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο τη Επιτροπή μα. Αυτό είπα προηγουμένω. I have a problem with Polish language. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εντάξει είμαστε. Okay. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει τώρα. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε. Θέλει κανείς το λόγο για την επίσκεψη στις Αζόρες. Όχι, οπότε να ευχαριστήσω και πάλι τους διοργανωτές της επίσκεψης αυτής. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή αποστολή και πολύ θερμή η φιλοξενία σε όλα τα επίπεδα στις Αζόρες. Είχαμε πολλές συνομιλίες και συναντήσεις με εκπροσώπους συνεταιρισμών, με παραγωγούς. Την έκθεση θα τη στείλουμε στην Επιτροπή, ώστε να λάβει γνώση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κατάστασης και των ε, θέσεων της Επιτροπής Άγκρη για το θέμα αυτό. Και μάλιστα πριν να στείλουμε επισήμω την έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τη στείλω στα μέλη της αντιπροσωπείας ε, για να την ελέγξουν. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι θερμά τους συναδέλφους για τη διοργάνωση αυτής της πολύ χρήσιμης ε, αποστολής της Αζόρες. Ήδη σας έστειλα και σε ευχαριστίες, αλλά δεν βλάπτει να τις επαναλαμβάνουμε και προφορικά. Και ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Στα έκτακτα αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την Τινησία. Η συντάκτρια της γνωμοδότης είναι η κυρία Γιλέρα Γκαρσία. Επειδή η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ανέβαλε την σχετική της ψηφοφορία και εμείς αναβάλουμε την ψηφοφορία της γνωμοδότησής μας για τις 11 Ιανουαρίου. Αλλά σήμερα μπορούμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Έγιναν συναντήσεις και με τους κερδισήγητες. Θα μας ενημερώσει σχετικά η συντάκτρια της γνωμοδότησης, η κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, ζητήσαμε αναβολή της ψηφοφορίας, γιατί στη συνάντηση που είχαμε τους κοιόδη ηγητέ, κρίναμε ότι καλό είναι να περιμένουμε τη μετάφραση των τροπολογιών πρώτα. Γι' αυτό και πρότεινα αναβολή της, ε, της ψηφοφορίας για την πρώτη μας συνεδρίαση του νέου έτους. Ήδη είχαμε μια πρώτη συνάντηση με τους και ηγητές στο Στρασβούργο και θα ήθελα να πω εν, εντόνως γιατί με ενδιαφέρει η γνώμη των συναδέλφων, ότι κατατέθηκαν 54 τροπολογίες, μερικές από συναδέλφους και ομάδες με πρόταση απόρριψης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διεύρυνση κατά 35.000 τόνους παράτασης ε, ε, και παράταση για διετία αυτής της ε, αύξησης ποσότητας ελαιολάδου από την Τινησία. Επίσης ζητήθηκε να διευκρινιστεί η προέλευση του ελαιολάδου, να έχει όντως παραχθεί στην Τινησία. Και άλλες τροπολογίες ζητούν μείωση αυτής της ποσότητας, Γιατί η ποσόστοση που ήδη ισχύει για την Τινησία, που είναι 56.000 τόνοι, είναι αρκετά μεγάλη, γιατί με εξαίρεση μία χρονιά δεν εξαντλήθηκε καν η ποσόστοση πριν την αύξησή της. Αυτό, αυτό λοιπόν είναι το αντικείμενο των τροπολογιών, η ποσότητα, η έκδοση των πιστοποιητικών ή η ύπαρξη εχεγγύων, ότι δεν θα μονιμοποιηθεί αυτή η αύξηση της ποσόστοσης. Αλλά θα παραμείνουμε στη διετή παράταση. Για να μην ξαναχρησιμοποιηθεί η γεωργία και τα γεωργικά προϊόντα, ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή, το ελαιόλαδο, ως αντάλλαγμα ή καλυμμένη ενίσχυση προς τη χώρα αυτή που έχει υποφέρει πολλά από τις δρομοκρατικέ επιθέσεις και από τις τελευταίες εξελίξεις. Εγώ κατάγομαι από την Ανταλουσία που είναι περιοχή με παραγωγή ελαιολάδου και μας προβληματίζει η στρέβλωση που ίσως δημιουργηθεί με την αύξηση τη της στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης μερικές τροπολογίες ζητούν να γίνει μια μελέτη επιπτώσεων αυτής της αύξησης της ποσόστοσης ελαιολάδου της Τινησίας ε, για τον ευρωπαϊκό κλάδο παραγωγής ελαιολάδου. Αυτά και θα ακούσω τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών και των υπόλοιπων συναδέλφων. Και τέλος να πω ότι από ό,τι ξέρω από την εισηγήτρια της ε, έκθεσης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, είναι το δεν έχει καταθέσει ούτε μία τροπολογία για την έκθεση. Οπότε, καλό θα ήταν όποια γνώμη και αν διαμορφωθεί στην Επιτροπή Γεωργίας, τη δική μας, ε, να χαίρει ευρείας υποστήριξη από τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Εράς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια της γνωμοδότησης για το έργο της και επίση ε, να ευχαριστήσω του συναδέλφου ε, του και την κυρία Γιούσου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά μια αύξηση, έκτακτη αύξηση για διετία της ποσότητας ελαιολάδου από την Τινησία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν είμαστε κατά καταρχήν, αλλά χρησιμοποιείται η γεωργία για την, για την ενίσχυση εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαμε στην περίπτωση της Ρωσίας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Άλλωστε, η κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Γεωργία αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι επιτρέπει στην εξωτερική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κατάχρηση τη γεωργία μα ή τη κτηνοτροφία μα ε, και να τις χρησιμοποιεί για την εξωτερική της πολιτική. Επίσης ε, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτή τη στιγμή η κοινοτική αγορά ελαιολάδου έχει χαμηλό επίπεδο ενισχύσεων. Οπότε για το 2016 θα μπορούσε να απορροφήσει την επιπλέον ποσόστοση. Αλλά αγνοούμε τι θα γίνει του χρόνου, το 2010, σε δύο χρόνια. Το 2017 δεν μπορούμε να προβλέψουμε, δεν είμαστε medium για να προβλέψουμε τις εξελίξεις. Οπότε είναι κάπως επικίνδυνη η παράταση για διετία. Γιατί για την πρώτη χρονιά γνωρίζουμε ότι μπορούμε να το να απορροφήσουμε την ποσότητα Για τη δεύτερη όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ε, χρειαζόμαστε και μια μελέτη επιπτώσεων για να δούμε ποιε θα είναι οι μελλοντικέ συνθήκε στον τομέα του ελαιολάδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για το 2016 35.000 τόνους και μετά να κάνει μια μελέτη και να δει κατά πόσο δικαιολογείται και για το 2017 η συνέχιση αυτή της ε, επιπλέον ποσόστοσης. Γιατί για να προτείνει για διετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την παράταση σημαίνει ότι έχει στοιχεία που ο ίδιος ο κλάδος ε, δεν διαθέτει για να δικαιολογεί αυτή την παράταση. Επίσης θα πρέπει να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις συνέπειες των μέτρων που προτείνεται και για το 2017. Αυτό θα ήθελα να μας σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, εν μία νυχτή δίνουμε στην Τινησία έκτακτη ποσόσταση που αυξάνει σχεδόν κατά 50% την ισχύουσα ποσόστοση. Γιατί 35.000 τόνοι ετησίως δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Επίσης έχουμε διμερεί συμφωνίες, διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την, Τινησία. Ίσως η ποσόστοση αυτή και η παράτασή της ερμηνευθεί εσφαλμένα ως πολιτική χειρονομία που θα έχει κάποια χρονική διάρκεια μπορεί η Τινησία να θεωρήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να διονύσει αυτή την παράταση της ποσόστοσης στη ε, Σύμφωνη Ελεύθερων Συναλλαγών που θα έχει με την, Τινησία. Οπότε αυτή η έκτακτη ποσόστοση καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προηγούμενο στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Τινησία για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Επίσης, ε, η νέα ποσόστοση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα μηχανισμό προστασίας για να αποφευθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και ρήτρα διασφάλιση σε περίπτωση που δημιουργηθεί τέτοια στρέβλωση ανταγωνισμού. Και μία ακόμη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απλουστεύσει τη μηνιαία διαχείριση και να τη μετατρέψει σε ετήσια διαχείριση. Δεν κατάλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η υποτιθέμενη απλούστευση ενέχει σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να αλλάξει ριζικά την ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καν δυνατότητα άμεση αντίδρασης. Δυστυχώς πρέπει να φύγω και δεν θα ακούσω την υπόλοιπη συζήτηση, αλλά περιμένω τις απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να φύγω να πάω τώρα σε άλλη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ να τηρείτε ο καθένας το χρόνο του, γιατί έχουμε μείνει ήδη πίσω. Ο κύριος Σελίμοβιτ. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους άλλους που συμμετείχαν στην ε, εργασία αυτή και που ήταν μεγάλη και σημαντική εργασία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να υποστορίξουμε τις συμβαστικέ τροπολογίες που προτείνει η συγκήτρια και άλλοι και θα προσπαθήσω να εξηγήσω πολύ σύντομα. Εξετάζοντας τα νούμερα, τι σημαίνουν τα νούμερα αυτά για τους τινήσιους και τι σημαίνουν για μας. Για τους τινήσιους όπως γνωρίζετε μετά από την τρομοκρατική επίθεση όλη η οικονομία τους έχει βυθιστεί. 15%, 15 της παραγωγής τους, δηλαδή έχει μειωθεί στο 15% η παραγωγή τους από το σύνολο που παρήγαν. Δίνοντας την ποσόστοση αυτή τους επιτρέπουν να διπλασιάσουν την παραγωγή τους. Δηλαδή μπορεί να φτάσουν μέχρι το 30% των όσων παρήγαν. Αυτό βεβαίω είναι τεράστια σημασία για τους ίδιου και τελικώ αυτό είναι και το ζητούμενο. Αλλά τι σημαίνει για μας? Η δική μας η παραγωγή έχει κατέβει 50%. 50%. 50% λοιπόν έχει μειωθεί η παραγωγή ολαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατανάλωση δε παραμένει περίπου στα ίδια. Λίγο έχει κατέβει. Τι σημαίνει λοιπόν 1% παραπάνω ελαιόλαδο που θα έρθει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάσαμε εμεί 50% τη παραγωγή και εισάγουμε 1%. Δεν μου φαίνεται λοιπόν κάτι τέτοιο να μπορεί να καταστρέψει την ευρωπαϊκή παραγωγή ελαιολάδου. Ελάχιστα πράγματα σημαίνει. Μιλάμε για δύο μεγάλες Ιταλικές πόλεις δηλαδή την παραγωγή, την αιτήσια την μάλλον κατανάλωση δύο μεγάλων τελικών πόλεων. Ενώ για τους Τινήσιους, όπως είπα, έχει τεράστια σημασία. Άρα δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την αποδυνάμωση της πρότασης της Κομισιόν που τη βρίσκω καλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ με την Άλντε και η δική μας πολιτική ομάδα θεωρεί ότι το μέτρο είναι προσωρινό, μπορεί μια χαρά να το απορροφήσει η αγορά μας και βεβαίως είναι τεράστια σημασία για την νησιακή οικονομία. Όπως είπα και στην Επιτροπή Εξωτερικών, για να αποφύγουμε τους κινδύνους να αποσταθεροποιηθούν οι αραβικές χώρες, αυτό δεν είναι βεβαίως ε, δεν είναι λάθο. Δεν είναι απάντηση και ούτε η γεωργία βεβαίω πρέπει να είναι η ηφηγένεια που θα θυσιαστεί στο βωμό της εξωτερικής πολιτικής. Σωστό αυτό που είπε κάποιο προηγουμένω. Όμω αυτό πρέπει να εξεταστεί ω θέμα από μόνο του. Γίνονται διαπραγματεύσει με την Τινησία και μέσα στι διαπραγματεύσεις αυτέ αυτό είναι ένα μικρό, μικρή σημασία στοιχείο. Άρα με τον τρόπο αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε την ε, πρώτη τροπολογία. Δεχόμαστε άλλες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για ε, εγγυήσεις για τους Ευρωπαίους Γεωργούς. Αυτά είναι λογικά πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω το μέτρο είναι προσωρινό τεχνικού χαρακτήρα που έχει όμως πολύ μεγάλη πολιτική σημασία και δεν αποτελεί διόλου προηγούμενο για το μέλλον. Ούτε μας κάνει να αποκλίνουμε από την πορεία μας. Θα βοηθήσουμε να αποκατασταθεί ένα μέρος της ε, τινησιακής οικονομίας, να σταθεροποιηθούν δουλειές και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Να βάλουν λοιπόν τα ευρύτερα συμφέροντα οι συνάδελφοί μας πάνω από τα πολύ στενά συμφέροντα που ενδεχομένως εκπροσωπούν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, υποστηρίζω πρώτα απ' όλα το έργο της συναδέλφου Αγγιλέρα και συμφωνώ κατά πολύ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Εράντς Καρσία. Θέλω πιο γενικά να μιλήσω. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό το ειδικό μέτρο για το παρθένο ελαιόλαδο είναι χρήσιμο πραγματικά για την Τινησία. Το θέτω σαν ερώτηση. Αναφισβήτα πρέπει να βοηθήσουμε την Τινησία. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν συζητούμε. Δέχτηκε την επίθεση τρομοκρατική, κατάρρευση η ε, παραγωγή. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να προσέξουμε. Μιλάμε για ένα μέτρο που θα καταλήξει να ευνοήσει μόνο κάποιου βιομηχανικού παραγωγού Ευρωπαίου που θα εισάγουν ε, το ελαιόλαδο την Ισία και μετά θα το μεταπίσουν και θα το πουλήσουν στην Ισπανία και την Ιταλία. Δημιουργούμε ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Σήμερα είναι το ελαιόλαδο για την Ισία. μετά θα βοηθήσουμε για να ευνοήσουμε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Δεν θα πρέπει η γεωργία ούτε αυτέ οι παραχωρήσει να είναι μονομερεί και να φορούν ένα μόνο προϊόν. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε την Τινησία και να δώσουμε τη δυνατότητα στι Τινησιακέ επιχειρήσει να αναπτυχθούν. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμη αυτή η αναβολή για τον Ιανουάριο. Θα μπορέσουμε να σκεφτούμε καλύτερα αυτό που κάνουμε. Δεν έχουμε εκτίμηση αντικτύπου. Είναι σημαντικά, σημαντικές οι ποσότητε, γιατί μιλάμε για διπλασιασμό τη ποσόστοση που υπήρχε πριν και δεν έχει χρησιμοποιήσει καν η Ισία. Δεν ισχύουν αυτά που έλεγε ο Σελίμοβιτ. Μιλάμε για έναν αντίκτυπο όσον αφορά την παραγωγή που δεν είναι ε, κοινό αντίκτυπο, εκτό αν κρύβεται πίσω από αυτό. Ίσως να υπάρχουν ευρωπαϊκά συμφέροντα και όχι την Ισιακά που θέλουν να καταφτάσει αυτό το ελαιόλαδο και μετά να το μεταπίσουν. Εγώ θα περίμενα... Ε, θα ήθελα πραγματικά να αναβληθεί για να μπορέσουμε να το, να το εξετάσουμε το θέμα. Παρακαλώ πιο σύντομη, γιατί μένουμε όλο και πιο πολύ πίσω στο χρόνο μας. Η κυρία Σένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ κατέθεσα τροπολογία για απόρριψη της πρότασης. Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου επικαλείται την αλληλεγγύη για να λάβει ένα μέτρο εμπορικής πολιτικής, ε, μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά. Θα ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιον θα ωφελήσει αυτό το μέτρο. Θα ωφελήσει όντως τα λαϊκά στρώματα, τους ε, αγρότες της Τινησίας ή μήπως θα ευνοήσει τον κλάδο ελαιολάδου γενικώ και όχι τους μικροπαραγωγούς. Σε τελική ανάλυση το μέτρο μήπως ε, προτείνεται για να μειωθεί η τιμή του ελαιολάδου, ώστε οι μεγάλες ε, βιομηχανίες της Ευρώπης να μπορούν να αγοράζουν φθηνό ελαιόλαδο, πλήττοντας έτσι τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Και τέλος, διαρωτώ με, πού είναι η μελέτη επιπτώσεων. Δεν θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί μελέτη επιπτώσεων για να λάβει η Επιτροπή μια τέτοια απόφαση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικότατη. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, τη στηρίζω, είναι καλή η έκθεσή της και εξίσου καλές είναι οι συμβαστικέ τροπολογίε. Όντω, όπως είπε ο κύριος Δεκάστρο, ε, κάνουμε πάλι ένα δώρο ε, εις βάρος των γεωργών με ξένα κόλληβα. Το πρόβλημα της Τινησίας εξαιτία των τρομοκρατικών επιθέσεων δεν είναι στο ελαιόλαδο, αλλά στον τουρισμό. Και εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα, με τα μέτρα για το ελαιόλαδο θα ευνοήσουμε τις ε, εταιρείε εισαγωγή που αγοράζουν φθηνό ελαιόλαδο και το πουλάνε και τις εταιρείε εξαγωγή της Τινησίας που έχουν πολύ γνωστά ονόματα. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Να πω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαμε την Αραβική Άνοιξη και όλοι είχαν ενθουσιαστεί γι' αυτό. Εγώ ήμουν κάπως διστακτικός. Αλλά το καλό ήταν ότι την Ισία δεν τα πήγε και τόσο άσχημα όσο οι άλλες αραβικές χώρες. Πραγματικά θα πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα για αυτούς να μας προμηθεύσουν με το προϊόν. Μου είπε ο Υπουργός της Τινησίας ότι είτε μπορούμε να σας παραδίνουμε προϊόντα, είτε τελικά θα έρθει ο κόσμος, θα έρθει ο λαός μας στις ακτές σας. Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες σε κάποιο βαθμό. Όπως είπε και κάποιος συνάδελφος, δεν τα συζητάμε αυτά τα θέματα τόσο πολύ, αυτό που συζητούμε το μέτρο δεν θα έχει τόσο φοβερό αντίκτυπο στην αγορά μας. Και τελικά θα χρειαστούν και χρόνο για να φτάσουν σε αυτές τις ποσότητες ή την ίσια. Στους δώσουμε όμω τη δυνατότητα να μας ε, προμηθεύσουν τα, με τα αγαθά τους. Κύριος Δικάστρο και άλλοι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν στην παραγωγή ελαιολάδου και πώς πάει η παραγωγή ελαιολάδου, νομίζω ότι αυτή η αύξηση του 1% θα ήταν ένα ευπρόσδεκτο μέτρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε να απορριφθεί αυτό το μέτρο που δεν βοηθά καθόλου τη Γεωργία ε, στην Ευρώπη, κυρίως κάποιες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Εγώ διαφωνώ απόλυτα με εκείνον που λέει αυτό το μέτρο δεν θα έχει κάποιο αντίκτυπο όσον αφορά την οικονομία μας. Θα έχει και πολύ μάλιστα. Και πώς. Διότι ε, λοιπόν, θα έχει, διότι η έλεγχη, αν είναι αιτήσιοι και όχι μηνιαίοι όπως ζητούμε, δεν θα μας επιτρέψουμε να αντιδράσουμε γρήγορα, ούτω ώστε να διορθώσουμε την κατάσταση. Θα έχει αντίκτυπο, διότι δεν θα έχει υπάρξει αντίκτυπος μόνο σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Διότι αυτό το μέτρο, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα ευνοήσει πάνω απ' όλα τις μεγάλους παραγωγούς που προφανώς θα αναμίξουν το δικό τους ε, λάδι με το φθηνό λάδι και θα θέσουν στην ευρωπαϊκή αγορά ένα προϊόν ακόμα ε, πιο φθηνό και αυτό θα βλάψει τους μικρούς παραγωγούς και τους καταναλωτές που δεν θα αγοράσουν ένα προϊόν και δεν θα έχει βέβαια προέλευση αυτό το προϊόν. Αυτού του είδους ε, η πρόταση θα πρέπει να απολυθεί. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, γιατί τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για τις διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν για την πρόταση αυτή και ευχαριστούμε και τις 54 τροπολογίες. Διαπιστώνουμε ότι υποστηρίζει η Επιτροπή την πρόταση αλλά θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση που αφορά τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Αυτή είναι και δική μας πρόθεση, σας διαβεβαιώ. Θα ήθελα να επενθυμίσω κάποια στοιχεία που είναι σημαντικά για να έχουμε σωστή προοπτική για την επίπτωση του μέτρου και να μην θεωρούμε ότι είναι διαβολικό μέτρο. Ε, λέμε ότι είναι ένα μέτρο προσωρινό πρώτα απ' όλα που θα εφαρμοστεί για δύο περιόδους, δύο περιόδους και η νέα ποσόστοση που δημιουργείται θα είναι διαθέσιμη από τη στιγμή που η παρούσα ποσόστοση των 56.500 τόνων που υπάρχουν στα πλαίσια του Συμφώνου Σύνδεσης ε, εξαντληθεί. Λοιπόν, εάν δεν εξαντληθεί αυτή η αρχική ποσόστοση δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθεί η νέα ποσότητα. Και τρίτο στοιχείο που θέλω να αναφέρω αυτό το μέτρο δεν προδικάζει και το αποτέλεσμα μελλοντικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια των, ε, της πλήρους συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών που θα διαπραγματευτούμε με την Τινησία. Τώρα όγκος αυτός 35.000 τόνοι μπορεί να φαίνεται μεγάλη ποσότητα σε σύγκριση με 56.500 τόνους που έχουμε στην παρούσα ποσόστοση αλλά η ανάλυση μας μας καταδεικνύει ότι μπορούμε να προτείνουμε αυτό τον όγκο ε, διότι δεν θεωρούμε ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο που θα διετάρασε την ευρωπαϊκή παραγωγή και τις ε, τιμές του ελαιολάδου στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή, αυτή 35.000 τόνοι είναι μόλις το 1,7% της παραγωγής ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για αυτή την ε, σοδιά, για αυτή την περίοδο και κατά την άποψή μας αυτός ο όγκος, αυτή η ποσότητα δεν θα διαταράξει τις τιμές του ελαιολάδου στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά περισσότερο οι διακυμάνσεις παραγωγής μπορούν να το κάνουν αυτό. Στην ευρωπαϊκή αγορά να επισημάνω λοιπόν ότι ήδη εκ των πραγμάτων σήμερα εισάγουμε από την Τινησία κατά μέσο όρο όταν βλέπουμε τις τελευταίες πέντε περιόδους βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισάγει λίγο πολύ κάθε χρόνο από την Τινησία περίπου 87.400 τόνους. Όσον αφορά αυτή την ποσότητα, πάνω από το μισό της ποσότητας, περίπου 40.000 τόνοι, εισάγονται στα πλαίσια της παρούσης ποσοστό στα πλαίσια της συμφωνία σύνδεσης και το άλλο ποσοστό, το άλλο μερίδιο εισάγεται μέσω του καθεστώτος της ενεργού τελειοποίησεως στο, σε αυτό το καθεστώς υπενθυμίζω ότι αυτός ο τελειωνιακός μηχανισμός επιτρέπει σε μια χώρα να εξάγει ένα προϊόν που υπόκειται σε μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επανεξάγεται εν συνεχεία προς τρίτη χώρα. Δεν υπόκειται λοιπόν σε τελωνιακό δασμό και αυτή είναι η πρακτική που ακολουθείται σήμερα. Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Η αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρειάζεται το ελαιόλαδο της Τινησίας ούτως ώστε εν μέρη να το μεταπεί και να το εμ, αποστέλει σε άλλους προορισμούς. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ποσότητα η νέα, οι 35.000 τόνοι θα αντικαταστήσουν το ποσό που εξάγεται μέσω της ενεργητικής μεταποίησης, αυτού που εξάγεται από την ενεργητική μεταποίηση, από αυτό το μηχανισμό. Άρα δεν θα υπάρξει ε, πρόσθετη ποσότητα ουσιαστικά. Και διαρωτώ γιατί ε, έχουμε διαρωτάστε γιατί έχουμε εξαντλήσει τα μηνύα όρια. Αυτά τα όρια είχαν καταρτιστεί για να περιορίζονται οι εισαγωγέ κατά του κρίσιμου μήνε, αυτού που ακολουθούν τη στιγμή της παραγωγή Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά αυτό το μέτρο δεν επέτρεψε να πετύχουμε το στόχο του περιορισμού των εισαγωγών ακριβώ αυτή την περίοδο, διότι τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου όταν, όταν ήταν πολύ χαμηλά τα όρια, οι ποσότητε ήταν μεγάλε διότι γινόταν εισαγωγή μεταξύ του καθεστώτος της ενεργού ε, τελειοποίησεως. Θεωρήσαμε ότι δεν ήταν χρήσιμο να παραμείνει αυτό το σύστημα και τέλος Α, δεν έχω πολλά να πω, τελειώνω. Όσον αφορά τη μελλοντική παραγωγή για τις επόμενες οδιές, η παραγωγή του τυνισιακού ελιδιού υπολογίζεται σε 170.000 τόνους. Οπότε δεν, είναι, δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση. Οι τροπολογίες δεν δέχεται τις τροπολογίες που απαιτούν την απόρριψη του κειμένου ή τη μείωση της προτινόμενης ποσότητας ή τη διάρκεια του μέτρου. Οι τροπολογίες που μιλάνε για κάποια μέτρα αποζημίωση των, Ευρωπα... των Ευρωπαίων παραγωγών νομίζω ότι δεν έχουν ε, θέση στην ε, πρόταση του κανονισμού, διότι δεν είναι αντικείμενο του κανονισμού να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα. Τέλος, θεωρούμε θετικές τις τροπολογίες που μιλάνε για μελέτη αντικτύπου. Θα πρέπει να αναλύσουμε δελεχέστερα τις σχετικές τροπολογίες, βέβαια επαγρυπνώντας και προσέχοντας τη διατύπωση, διότι είναι σαφές ότι η κατάσταση της αγοράς του ελαιολάδου υπόκειται στην επίδραση και άλλων παραγόντων, πολλών παραγόντων πέραν των εισαγωγών από την Τινησία. Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει σωστό συσχετισμός των παραγόντων για να μην φορτώσουμε σε αυτές τις ε, μέτριου μεγέθους εισαγωγής από την Τινησία όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του ελαιολάδου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ήταν ε, εκτενέστατη συζήτηση και έχουμε μείνει πίσω. Σας ε, παρακαλώ. Μια και θα ψηφίσουμε στις 11 Ιανουαρίου έχουμε χρόνο αλλά μην περιμένετε άλλο για να καταθέσετε τις τροπολογίες σας ώστε μέχρι το Δεκέμβριο οι συγγήτρια και οι σκιώδεις συγγητές να μπορέσουν να εξετάσουν το θέμα και να μας προετοιμάσουν για την ψηφοφορία. Παρακαλώ τη συντάκτρια της γνωμοδότησης, αλλά πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Όντως, δύο λόγια μόνο για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και ηγητές και τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να πετύχουμε στο μέτρο του δυνατού μια συνένεση στην Επιτροπή Γεωργίας και να πω ότι όλα έχουν αντίκτυπο στο, στον τομέα του ελαιολάδου. Ε, προηγουμένως ήταν 4 ευρώ το κιλό το, ελαιό, το λίτρο το ελαιόλαδο τώρα είναι 2,55. Έχει ήδη μειωθεί η τιμή ελαιολάδου δηλαδή. Μην νομίζετε ότι αυτό το μέτρο δεν επιδρά στην, στον προσδιορισμό της τιμής. Πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε πριν τα Χριστούγεννα να ολοκληρώσουμε τη σύνταξη της γνωμοδότησης και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε κανονικά τον Ιανουάριο όπως έχουμε προγραμματίσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπερνάρ Βαλά, που είναι Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων. Θα... Μην ξεχνάτε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων είναι για τα ζώα ό,τι είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την Υγεία των Ανθρώπων. Παρακαλώ λοιπόν τον Γενικό Διευθυντή να λάβει θέση. Ο κύριος Βαλάτ ε, είναι εμπειρογνώμονας, ε, παίων στα θέματα αυτά. Εδώ και πολλά χρόνια Γενικό Διευθυντή ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων. Έχει πάρα πολλά προσόντα. Είναι κορυφαίος εμπειρογνώμονας, οπότε θα μας διαφωτίσει για θέματα που μας είναι και πολύ ενδιαφέροντα και άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Θα μιλήσει για, τα, για τη μικροβιακή αντοχή, για το πρόβλημα που έχουμε με την πανόλη των χείρων, για την υγεία των ζώων. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων μαζί σας κύριε Γενικέ. Και περιμένουμε την ενημέρωση για το τεράστιο έργο που πραγματοποιεί ο οργανισμός σας. Merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τιμή για μένα και για τον οργανισμό μας να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες μας και τα θέματα τα σημαντικά που αφορούν την υγεία και την ευημερία των ζώων στον πλανήτη μας. Θα παρουσιάσω PowerPoint, έχω μια παρουσίαση PowerPoint για να δείτε καλύτερα το θέμα. Έφερα και πολλά έγγραφα που βρίσκονται επί τάπητος, ε, στο τραπέζι μάλλον δεξιά μου, που μπορούν να τα συμβουλευτούν και να τα πάρουν όλοι οι βουλευτές αυτά τα έγγραφα. Αν είχατε την καλοσύνη να δείξετε τη διαφάνεια στην οθόνη. Σας ευχαριστώ. Ο οργανισμός μας λοιπόν δημιουργήθηκε το 1924, πολύ πριν από τον ΟΗΕ και αυτό εξηγεί ότι είμαστε ανεξάρτητοι από το δίκτυο του ΟΗΕ και τα κράτη-μέλη μας είναι ικανοποιημένα από την κατάσταση αυτή. Το 2003 άλλαξε ε, η ονομασία από το Διεθνές Γραφείο των Επιζωτιών ε, μετονομάστηκε σε Παγκόσμιο Οργανισμό για την, ανθρώπινη, για την ε, Υγεία των Ζώων. Ε, είναι στο Παρίσι έδρα μας. Έχουμε 13 γραφεία στον κόσμο. Τα περισσότερα είναι στην Ευρώπη και θα συνεχίσω αργότερα σε λεπτομέρειες. Έχουμε 180 κράτη-μέλη. Μας λείπει η προσχώρηση κάποιων μικρών νησιών του Ειρηνικού και της Καραϊβικής που δεν έχουν ζώα στην πράξη ε, και θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου ε, παρουσιάζοντας τις μεγάλες αλλαγές, τις μεγάλες εξελίξεις ε, που αφορούν την κτηνιοτροφία, κινδύνους όσον αφορά την υγεία των ζώων και όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, τις μεγαλύτερες μετακινήσεις αγαθών και προσώπων, την αλλαγή του κλίματος που πολύ συχνά συνδέεται με τις παρεμβάσεις της ανθρωπογενής ε, δραστηριότητας του ανθρώπου και αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην παγκόσμια διάδοση των μικροβίων και των φορέων που ε, διευκολύνουν την μεταβίβαση των ασθενειών στον άνθρωπο και στα ζώα σε νέες γεωγραφικές ε, περιοχές και η Ευρώπη ιδιαίτερα πλήττεται και επηρεάζεται από τις εξελίξεις αυτές, κυρίως από ε, διάφορα μικρόβια που προέρχονται από την ε, Αφρική. Και αυτό έχει βέβαια και αντίκτυπο όσον αφορά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών της προλήψεως και του ελέγχου των διαφόρων ασθενειών των ζώων. Ε, στον κόσμο βλέπουμε ότι υπάρχει σχέση στενή μεταξύ των φτωχών περιοχών της Πέθρου και της ε, ιδιοκτησίας ζώων. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο φτωχοί άνθρωποι βασίζονται στο ζώο για να επιβιώσουν. Επίσης βλέπουμε ότι ε, το να έχει κανείς ένα ζώο είναι σημαντικό στάδιο για να μπορεί να ξεφύγει από τη φτώχεια. Και γι' αυτό η προστασία του κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου των φτωχών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις πολιτικές που αφορούν τη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, βλέπουμε επίσης ε, να αναδύονται και νέες οικονομικές δυνάμεις, νέες χώρες και στις χώρες αυτές αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μία μετακίνηση από το επίπεδο φτώχειας προς τη μεσαία τάξη και αυτό οδηγεί σε πάρα πολύ σημαντική κατανάλωση ζωικής, ζωικών πρωτεϊνών, γάλακτος, κρέατος. Λοιπόν, ενώ έχει, δεν αναπτύσσεται η κατανάλωση, δεν αυξάνεται στις αναπτυγμένες χώρες, εκεί εκθετικά ε, αυξάνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, οπότε συνολική κατανάλωση ε, ζωικών προϊόντων στον κόσμο ε, αυξάνεται με πολύ σημαντικούς ρυθμούς και αυτό έχει συνέπειες όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία και για τις αναπτυγμένες χώρες και αυτό θα πρέπει να έχει αντίκτυπο όσον αφορά τον καθορισμό των πολιτικών που ακολουθούν αναπτυγμένες χώρες όσον αφορά την πρόληψη. Να πω κάποια λόγια για τα πιο επίμαχα θέματα όσον αφορά το συσχετισμό ε, ανθρώπων και ζώων στον κόσμο, θετικές συνέπειες, αρνητικές συνέπειες της σχέσεως μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Υπάρχουν λοιπόν ε, διαφωνίες όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχουν τα ζώα, τα κιακά ζώα στο περιβάλλον. Είναι ένα θέμα περιπλοκότατο και έχουμε στοιχεία διαφορετικά που διατίθενται. Αν, αν τα δημοσιεύει η ΦΑΟ Φερρυπίν, το Livestock Shadow πρόσφατα ή σύμφωνα με αυτά που δημοσιεύονται από το ΖΙΕΚ ε, ανάλογα με τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των, ε, του αντιχτύπου και των συνεπειών που υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ε, το μήνυμά μας το βασικό λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην χάσουμε τα πάντα στα μέτρα που λαμβάνουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις θετικές πτυχές των ζώων να θυμηθούμε ότι το 1 τρίτο του πλανήτου δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε χωρίς τα μερικαστικά που αλλάζουν την ε, κυταρίνη ε, και άλλα φυσικά προϊόντα σε προϊόντα υψηλής ποιότητας διατροφικής που επιτρέπουν σε πληθυσμούς να επιβιώνουν δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η ζωική πρωτεΐνη παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κεφάλου των παιδιών και χωρίς αυτές τις πρωτεΐνες βλέπουμε να υπάρχουν προϊόντα ε, σοβαρά όσον αφορά την υγεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν την προσοχή ότι πρέπει να λάβουμε τις θετικές στοιχές της κτηνοτροφίας υπόψη όταν ε, συζητούμε τον αντίκτυπο που έχει αυτή στο περιβάλλον. Όσον αφορά τις διαφορές που υπάρχουν για την ανθρώπινη υγεία, τις απόψεις, τις διαφορετικές που υπάρχουν. Έχουμε παράδειγμα, μάθαμε, μια δημοσίευμα μιας οργανώσεως μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναφέρεται στον κίνδυνο υγείας που συνδέεται με την κατανάλωση μεταποιημένων ζωικών προϊόντων. Παραδείγματος χάρη τα αλλαντικά με πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά τη στάση τελικά των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο και παραδόξως αυτή η μελέτη συσχέτιζε την κατάσταση με το ερυθρό κρέας χωρίς όμως να δίνει επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τη διασύνδεση του κινδύνου με το ερυθρό κρέας. Ε, και αυτό πριν την COP21 δημοσιεύτηκε. Αυτού του είδους ε, οι θέσεις θα πρέπει να εξετάζονται με πάρα πολύ μεγάλη επιστημονική αυστηρότητα και είμαστε αντίθετοι, επαναστατούμε κατά πολύ ε, γρήγορων ε, ερμηνεών όσον αφορά επιστημονικές μελέτες. Υπάρχει και άλλη διαφορά όσον αφορά το κόστος του ελέγχου και της προλήψεως όσον αφορά τις ασθένειες, δηλαδή ε, της εισόδου ε, ασθενειών σε διάφορες ε, περιοχές που ήταν ακέραιες, δεν είχαν αυτή την ασθένεια. Και το κόστος που πρέπει να καταβληθεί για να εμποδιστεί να εισαχθούν κάποιες τέτοιες ασθένειες σε σύγκριση με την αντιμετώπιση κρίσεων που είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς προλήψεως και ανεπαρκών μέσων που διατίθενται. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται και αυτό σχετίζεται με ένα είδος ε, ε, του κόστου των ασφαλιστικών, των μέτρων για την ασφάλεια που λαμβάνουν τα μέτρα. Αυτοί οι οικονομικοί υπολογισμοί που κάναμε και εμείς πάντα οδηγούν στο να συμπεραίνουμε ότι το κόστος της εποπτείας ε, είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος αντιμετωπίσεως μιας κρίσης άμα ξεσπάσει. δεν κλείνουμε τα, τους πυροσβεστικούς ε, σταθμούς γιατί ε, δεν υπήρχαν βροχές, δεν έπεσε νερό κλπ. Λοιπόν τώρα όσον αφορά την εξολόθρευση ζώων όταν ξεσπάσει μια επιζωοτία υπάρχουν θέματα, υπάρχει ισχυρή αντίδραση όταν αυτές ε, όταν σφάζονται πολλά ζώα, όταν έχουν ασθενήσει. Εμεί είμαστε επιφορτισμένοι με το να καθορίσουμε τι μεθόδου καταπολέμηση ασθενειών. Η πολιτική του οργανισμού μα είναι πάντα να δίνουν προτεραιότητα στην χρήση του εμβολιασμού. Δυστυχώ υπάρχουν περιπτώσει όπου δεν μπορούμε να απαλλαχθούμε από μια ασθένεια χωρί να εξοντώσουμε κάποια άρρωστα ζώα, όπως ε, στην περίπτωση της γρήπη των πτηνών ε, χρειάζεται να υπάρχει σωστή επικοινωνία με τους ε, πολίτες μας, να μπορούμε να εξηγούμε στους πολίτες ότι θα πρέπει στο μέγιστο βαθμό να μειώσουμε τον αριθμό των ζώων που εξολοθρεύονται, αλλά σε εξαιρετικές περιστάσεις η προστασία της δημοσίας υγείας είναι αυτή που υπερισχύει και έχει προτεραιότητα. Λοιπόν, έναντι αυτών των διαφορών, των επιμάχων ζητημάτων, ε, ποια η συνεισφορά του οργανισμού μας όσον αφορά τη διεθνή κοινότητα, ε, είμαστε ένας διακυβερνητικός φορέας, ένας οργανισμός διακυβερνητικός και καθορίζουμε τις μεθόδους ελέγχου των ζωονόσων και των μεταδοτικών αυτών. 60% των ανθρωπίνων ασθενειών έχουν ζωική προέλευση. Επιτιθέμενοι στην πηγή, λοιπόν, στις ζωονόσους, προστατεύουμε την ε, ανθρώπινη υγεία, τη, τη δημόσια υγεία. Οι προδιαγραφές μας υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη δημοκρατικά και αναγνωρίζονται από το ΠΟΕ. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα και στη διεθέτηση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των χωρών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους ζωικά προϊόντα. Είμαστε μόνος ο οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει, είναι εντολοδόχος και ε, όσον αφορά την υιοθέτηση προδιαγραφών για την ευημερία των ζώων. Μπορούμε να αποφασίζουμε από αυτού. Έχουμε ήδη από το 2004 εθετήσει πολλά, πολλά, πολλά τέτοια μέτρα. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα που είναι σημαντικότατο για την Επιτροπή σας. Το γνωρίζω αυτό. Έχουμε επίσης την ευθύνη να δημοσιεύουμε στοιχεία για την παγκόσμια κατάσταση αφορά τις ασθένειες στα κράτη-μέλη μας και διαχειριζόμαστε ένα σύστημα που αποκαλείται WAHIS, Έχουμε 180 χώρες που συνδέονται με ε, τον σερβερ μας, με τον υπολογιστή μας και διαχέουμε τις πληροφορίες στο κοινό μέσω ιστοσελίδας. Έχω φέρει μια, ένα μικρό βίντεο, ένα CD-ROM που είναι εδώ στο τραπέζι, είναι πολύ σύντομο και σας ενημερώνει όσον αφορά τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι χώρες, όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με την κατάσταση που κρατεί στη χώρα τους σχετικά με τις ζωονόσους και έχουμε συμφωνία με το Κόντεξ Αλιμεντάριους ούτως ώστε οι προδιαγραφές που καταρτίζουμε όσον αφορά ε, την ε, διατροφή να μην ε, είναι αντιφατικές, να μην δημιουργούν κενά και γι' αυτό ασχολούμαστε με προδιαγραφές μέχρι την έξοδο από την εκμετάλλευση και ο κόντεξ αλιμεντάριος ασχολείται με προδιαγραφές που αφορούν τα τρόφιμα μετά την έξοδο από την φάση της ε, παραγωγής του τροφίμου. Λοιπόν, τώρα οι προδιαγραφές που ετοιμάζουμε και εγκρίνουμε αφορούν τα συστήματα ενημέρωσης πληροφοριών όσον αφορά τις ασθενείες κατά κάτω μέλος, τρόποι πρόληψης και ελέγχου των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης και της ποιότητας των δοκιμών, των διαγνωστικών και των εμβολίων, και ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τα προϊόντα και τα, και τα προϊόντα ζωικής και των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, ποιο διαγραφές πρέπει να εφαρμόζονται για να μην εισάγονται μικρόβια στην επικράτεια των χωρών που, που κάνουν τις αγωγές ε, χωρίς να χρησιμοποιούνται σαν πρόσχημα τα θέματα υγείας για προστατευτισμό χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις. Έχουμε και προδιαγραφές για την ευμερία των ζώων, για την ασφάλεια των προϊόντων ε, σε επίπεδο εκμεταλλεύσεως, για την ποιότητα των εθνικών συστημάτων για την υγεία των ζώων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Καλή λοιπόν διακυβέρνηση, καλή διαχείριση όσον αφορά τα θέματα υγείας στι χώρες μας Έχουμε λοιπόν σχετικέ προδιαγραφές για αυτή τη διακυβέρνηση και εκεί συμπεριλαμβάνεται και η ποιότητα της καταρτήσεως των κτηνιάτρων ε, στον κόσμο. Και τέλος εκπονούμε και προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση για θέματα υγείας που αφορά όλες τις αγωγέ προϊόντων ζώων ή προϊόντων ζωικής ε, προελεύσεως. Έχουμε και την αποστολή να αναγνωρίζουμε το καθεστώς όσον αφορά την υγεία των κρατών μελών μας έναντι διαφόρων πολύ σημαντικών ασθενειών. Ε, λοιπόν, όσον αφορά την ασθένεια της τρελής αγελάδας, όπου ε, ανήκε σε έναν κατάλογο, όπου εκεί ψηφίζουμε για να αποφασίσουμε αν κάποια χώρα ε, είναι ελεύθερη από την ασθένεια και έχουμε τις κατηγορίες Έχουμε την κατηγορία του απροσδιορίστου κινδύνου, δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση ή θεωρούμε ότι είναι αρνητική. Καθεστώς κινδύνου ελεγχομένου, δηλαδή η χώρα έχει εφαρμόσει όλα τα μέτρα που είναι αποδεκτά για να ελεγχθεί η ασθένεια αλλά δεν είναι σίγουρα ότι είναι ελεύθερη και μετά μελιτέως κίνδυνος που είναι η καλύτερη κατάσταση ε, όσον αφορά τις χώρες σχετικά με τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει αυτή η ασθένεια και αυτή η ταξινόμηση που υφετήθηκε από τη Γενική μας Συνέλευση είχε συνέπειες όπως αφορά την, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίσαμε τα περισσότερα κράτη-μέλη ότι είχαν θετική κατάσταση και αυτό είχε σημαντικότατες συνέπειες όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο των χωρών της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ενώσεως. Επίσης αναπτύσσουμε και την τον διαχωρισμό σε ζώνες, αυτή την έννοια, όταν υπάρχει μια ασθένεια σε μια χώρα, αντί να αποκλείουμε όλες τις εξαγωγές από αυτή τη χώρα, προβλέπουν οι κανόνες μας τη δυνατότητα να δημιουργείται μια μολυσμένη ζώνη από την οποία απαγορεύονται εξαγωγές, αλλά η υπόλοιπη χώρα μπορεί να συνεχίσει να εξάγει και ξέρετε ότι πρόσφατα οι Ηνωμένε Πολιτείε δέχτηκαν αυτή την έννοια ως, όσον αφορά τον αυτό των χείρων ε, και ως, ως χωρίς να πλήττεται ε, το εξωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, έχουμε και άλλη έννοια, μία ενιαία υγεία. Δηλαδή πώς να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με την υγεία των ζώων και εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη δημόσια υγεία και γι' αυτό συνήψαμε συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την ΦΑΟ και πήραμε σαν παράδειγμα, σαν προτεραιότητα την ΛΙΣΑ ε, και τη γρήπη των πτηνών, γρήπη των ζώων και την ε, αντίσταση στα μικρόβια που όπως ξέρετε είναι ένα θέμα που γίνεται όλο και πιο σημαντικό ε, στο θεματολόγιο όλων των ε, κυβερνήσεων, κυρίως όσον αφορά τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Θα επανέλθω από αυτών των θεμάτων, διότι θα παραθέσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορούν να σας προσελκύσουν την προσοχή. Έχουμε επίσης μαζί με τους εταίρους μας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ετοιμάσαμε και έναν οδηγό προς προσοχή όλων των χωρών μελών μας για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών των αρμοδίων την υγεία των ζώων και των υπηρεσιών των υπευθύνων για τη δημόσια υγεία. Εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος, το ζώο και το περιβάλλον όσον αφορά την πρόληψη του κινδύνου. Αυτός ο οδηγός επιτρέπει τη βελτίωση των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα αυτό και να βελτιωθεί η συνεργασία αυτή που γίνεται πολύ σημαντική σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποιημένο ε, και αλλαγών κλιματικών. Ιδού λοιπόν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα όσον αφορά τα διάφορα προϊόντα που σας ε, προανέφερα πώς δρούμε για να βελτιώσουμε την όλη διαχείριση και διακυβέρνηση των συστημάτων υγείας των ζώων στα κράτη-μέλη μας. Λοιπόν, έχουμε ένα μηχανισμό που επιτρέπει στα κράτη-μέλη μας να ζητήσουν μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του κατά πόσο συμμορφώνονται με τις ποιοτικέ προδιαγραφές των εθνικών συστημάτων. Έχουμε πάνω από 100 εμπειρογνώμονες που έχουν καταρτιστεί γι' αυτό και προβαίνουν στις αξιολογήσεις ε, ε, κατόπιν ετήσιος των χωρών. Και μετά όταν γίνει η διάγνωση όπως την αποκαλούμε, γίνεται αποδεκτή βέβαια αυτή από τη χώρα που αναγνωρίζει και τα διάφορα κενά που διαπιστώνονται και μπορούμε τότε να προτείνουμε στις χώρες Δηλαδή αποτιμούν το κόστος της συμμόρφωσης εμπειρογνώμονε με τις ποιοτικέ προδιαγραφές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για τις αναπτυγμένες χώρες ή τις χώρες εκείνες που θέλουν να στηρίξουν την ποιότητα των συστημάτων υγείας των φτωχών χωρών, διότι θεωρούν ότι αυτό είναι απειλή για εκείνες. Υπάρχει ένα πλαίσιο για προσανατολισμό των χρηματοδοτήσεων για να βοηθήσουν τις χώρες εκείνες που θέλουν συμμορφωθούν με τις παγκόσμιες ποιοτικές προδιαγραφές του συστήματος. Προτείνουμε και αυτό αφού εντοπίσουμε τα κενά, τα σημαντικά και τη θεραπεία, τη διόρθωση αν θέλετε. Προτείνουμε στις χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες όλες ιδιαίτερως μια άμεση στήριξη, τεχνογνωσία όσον αφορά την κτηνιατρική νομοθεσία για την συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα συστήματα υγείας και πρόληψης και ελέγχου των ασθενειών αυτό τους δίνουμε στήριξη όσον αφορά την, την, την μόρφωση στον τομέα, την παιδεία στον τομέα της ιατρικής, διότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουν πολιτική για την ε, υγεία των ζώων χωρίς να έχουμε καλά κατατισμένους κτηνιάτρους. Έχουμε 135 χώρες ε, που εμπλέκονται στο σύστημα και το, το Διεθνές Ταμείο Ανάπτυξης ε, ε, χρησιμοποιεί τα διάφορα προϊόντα χρηματοδίτησης για να βοηθά αυτές τις χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος δωρητής ε, σε αυτό το τομέα ε, μέσω Παγκοσμίου ε, Ταμείου που διαχειριζόμαστε μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις χώρες που το επιθυμούν. Παραδόξως τώρα έχουμε πλούσιες χώρες που μας ζητούν να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση για να μπορέσουν και αυτές να τοποθετηθούν εν συγκρίση με τις κυβερνήσεις τους για να δουν πόσο ποιοτικό είναι το σύστημά τους να έρθουν σε ένα διάλογο με τα κοινοβούλια τους ή την κυβέρνησή τους για τη βελτίωση της ποιότητας. Έχουμε την Αυστραλία, Φερρυπίν, έχουμε τον Καναδά, την Ιαπωνία, οι οποίες χώρες αξιολογούνται κατόπιν αιτήματός τους και συστήνω στις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δεν έχουν ακόμα κάνει τέτοιο, που δεν έχουν ζητήσει την ανεξάρτητη αξιολόγηση, έχουν κάνει αυτοαξιολόγηση, συστήνω στις χώρες λοιπόν να ζητήσουν να διεξαχθούν αυτές οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις ε, και βέβαια οι χώρες ε, είναι οι διοκτήτες αυτών των αξιολογήσεων. Δεν υπάρχουν αρνητικές ε, εμπορικές συνέπειες από την αξιολόγηση. Να πω κάποια πράγματα εν είδη παραδείγματος για το One Health, μια και μοναδική υγεία. Αυτή την έννοια που προανέφερα, σας την εξηγήσω. Λοιπόν, έχουμε επίσημη συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το ΦΑΟ για να μπορούμε από κοινού να δρούμε για να συντονιζόμαστε όσον αφορά την υγεία των ζώων και την δημόσια υγεία από κοινού και θέτοντας προτεραιότητες όσον αφορά τη γρήπη, τη λύσα και την αντίσταση στα μικρόβια. Γνωρίζετε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει διεθνή ε, κανονισμό για την υγεία που ψηφίζεται από όλα τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη υπο, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά την ποιότητα των συστημάτων τους δημοσίας υγείας. Ε, αυτό δεν αφορά μόνο το εσωτερικό των χωρών, αλλά αφορά και τον κίνδυνο που δημιουργούν αυτές οι χώρες για τον υπόλοιπο κόσμο όταν δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Λοιπόν, ε, έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος μηχανισμός επιτρέπει να εφαρμόζεται το δικό μας σύστημα αξιολόγησης της ορθής διακυβέρνησης που περιέγραψα και αυτόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ούτως ώστε τα δύο συστήματα να συγκλίνουν στο επίπεδο διεπαφής ανθρώπου, άνθρωπος ζώο ε, περιβάλλον και χρησιμοποιούμε και τον οδηγό που σας ε, παρουσίασα και σας ανέφερα. Ε, ήδη έχουμε δωρητές οι οποίοι επιδοτούν τις δράσεις μας στις φτωχότερες χώρες για να επιταχυνθεί το τρόπος η αύξηση της ποιότητας, η βελτίωση της ποιότητας του συστήματος που στατεύει την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. Εφαρμόζουμε επίσης και διάφορα προγράμματα για να υπάρχει, να πλησιάσει ο ιδιωτικός τομέας με το σύστημα της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, να υπάρχει συνεργασία των ιδιωτικών ε, ε, κτηνιάτρων με αυτούς του δημοσίου τομέα και να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των γεωργών, των κτηνοτρόφων ε, για τα θέματα αυτά και να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των ιδιωτικών κτηνιάτων και είναι σημαντικός ο ρόλος και των κτηνιάτων. Δημιουργούμε ένα τρίγωνο για να μπορούμε να εγγυηθούμε την πρόληψη των ασθενειών. Άλλο παράδειγμα, τα προγράμματά μας που εφαρμόζουμε για την κατάρτιση, για βελτίωση της, του δυναμικού που υπάρχει, των δυνατοτήτων που υπάρχουν στις χώρες. Ε, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες βοηθούμε, αλλά κυρίως ισχύουν αυτά και για όλες τις χώρες μέλη, διότι χρειάζεται να υπάρχει μια ανακύκλωση ενημέρωσης όσον αφορά τις μεθόδους πρόληψης, τις πιο νέες μεθόδους να μαθαίνουμε για την πρόληψη των νόσων. Διοργανώνουμε διασκέψεις σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου σε τριμήνο για τη συζήτηση των θεμάτων αυτών. του χρόνου στο Μεξικό θα γίνει μια μεγάλη παγκόσμια διάσκεψη για την προστασία των ζώων που θα εγκρίνει και σχετική στρατηγική. Εμείς προσφέρουμε σε όλες τις χώρες μια διαρκή ανακύκλωση ενός εθνικού εμπειρογνώμονα και συνομιλητών, δηλαδή focal points, στις ε, ε, χώρες για να συμβάλλουν στην προσπάθεια των όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις για να μπορούν να προβλέπουν τις επιπτώσεις των αποφάσεων στην ε, υγεία των ζώων. Και έχουμε focal points σε 180 χώρες για, τα, για τους τομείς θεμάτων όπου δραστηριοποιούμεθα. Και για να διασφαλίζουμε την ε, ποιότητα των κανόνων που προτείνουμε και εγκρίνουμε, έχουμε ένα δίκτυο 300 ε, εργαστηρίων ανά τον κόσμο υψηλού επίπεδου για την μελέτη των θεμάτων του αγώνα κατά των ζωονόσων. Και από αυτά ένα μεγάλος αριθμός βρίσκεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίζουν ουσιώδη ρόλο για την στήριξη του οργανισμού μας σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιούμεθα και πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις ε, μεγάλου κύρους. Δημοσιεύουμε επίσης και κατευθυντήριες γραμμές για την κτηνιατρική εκπαίδευση και έχουμε κατορθώσει να εναρμονίσουμε το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να εξασφαλίσουμε ώστε όλοι οι κτηνίατροι να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ε, εκπαιδεύσεως για την απόκτηση των ε, δεξιοτήτων που τους είναι απαραίτητες για να μπορούν να επιτελέσουν το έργο της προστασίας το, της υγείας των ζώων και βέβαια και του κοινού. Τώρα, λίγα για την ε, προστασία ή την ευημερία των ζώων. Έχουμε λάβει βεβαίω την εντολή να παράγουμε του ε, κανόνε, τα πρότυπα για την προστασία τη υγεία των ζώων. Πολύ σημαντική δραστηριότητα αυτή. Θα ήθελα επίση εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Όταν αρχίσαμε να φτιάχνουμε του κανόνε αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η μόνη περιοχή του κόσμου που επέβαλε στους επιχειρηματίες της είτε ε, αγρότες, είτε μεταποιητές, είτε οτιδήποτε άλλο, ε, δεσμευτικούς κανόνες για την ευημερία των ζώων. Και οι τρίτες χώρες, δύο οι μεγάλες παραγωγές και εξαγωγικές χώρες, δεν επέβαλαν τέτοιους ε, όρους στους παραγωγούς τους. Υπήρχε λοιπόν εκεί μια διαφορά ανταγωνιστικότητας που οφείλονταν στην εφαρμογή των δεσμευτικών αυτών κανόνων. Από τότε λοιπόν που ο οργανισμός μας παράγει κανόνες, πρότυπα και που ε, γίνονται σεβαστά όλο και περισσότερο και από τρίτες χώρες, δυστυχώς όχι από όλες αλλά όλο και περισσότερο, η διαφορά στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών παραγωγών και των παραγωγών τρίτων χωρών τίνει να μειώνεται σιγά αλλά σταθερά. Θα έλεγα τώρα ε, δυστυχώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ε, στις συμφωνίες του η αναγνώριση των κανόνων της ευημερίας των ζώων που παράγει ο εργατικός μας οργανισμός δεν είναι ξεκάθαρη, δεν αναφέρεται καν στην ε, συμφωνία για τα φυτοϊγειονομικά προϊόντα, ορισμένα άλλα στοιχεία των κανονισμών του ΓΚΑΤ επέτρεψαν πρόσφατα στη διάρκεια του πάνελ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά για ορισμένα προϊόντα φώκιας επέτρεψαν για πρώτη φορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να τοποθετηθεί επί ενός θέματος που έχει σχέση με θέματα ευημερία των ζώων, διότι εκεί τέθηκε θέμα του τρόπου ε, θανάτωσης των φωκών στον Καναδά και για πρώτη φορά λοιπόν Γι' αυτό λοιπόν εκεί βρισκόμαστε. Θέλω να πω όμως ότι ακόμα βρισκόμαστε μακράν συμφωνίας ε, με συνένεση στον ε, παγκόσμιο, ή μάλλον με ομοφωνία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για θέματα ευημερία των ζώων. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι οι κανόνες που έχουν γίνει δεκτοί από τις 180 χώρες μέλη μας ε, χρησιμοποιούνται από όλους τους διαπραγματευτές στις διμερείς διαπραγματεύσεις για ε, τις εμπορικές συμφωνίες και αποτελούν τη βάση για συμφωνίες και για συζητήσεις που οδηγούν σε συμφωνίες. Καμιά φορά φτάνουν μέχρι να περιληφθούν και στις συμφωνίες, πάντως είναι απαρέγκλητη βάση για τις συζητήσεις για τις μελλοντικέ ε, διμερείς ε, συμβάσεις. Άλλο παράδειγμα, οι τράπεζες, οι περιφερειακές τράπεζες εμβολίων για παράδειγμα για την Δύσα που ε, χτυπάει πολλούς ανθρώπους, πολλά εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, για την πανόλη των μυρικαστικών, μεγάλη ε, πληγή και απειλή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον αυτόδη πυρετό που εδώ όλοι γνωρίζετε καλά. Αυτές οι τράπεζες εμβολίων επιτρέπουν την επιλογή εμβολίων ε, υψηλής ποιότητας για να είναι εξασφαλισμένη η δράση τους, να είναι εγγυημένη η άμεση ε, προμήθειά τους εφόσον είναι απαραίτητο και είναι ανοιχτές οι τράπεζες, ε, εμβολίων είτε για να διαθέτουν δωρεάν σε πιο φτωχές χώρες τα εμβόλια είτε για να επιτρέπουν την εκκίνηση της παραγωγής εμβολίων από επιχειρήσεις, από ε, εταιρείε που θέλουν να συμβάλλουν σε εκστρατείες σε ορισμένε Και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην δημιουργία και στη λειτουργία αυτών των τραπεζών εμβολίων υπό ορισμένου όρου, αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Έρχομαι στο τελευταίο κεφάλαιο της ομιλίας μου. Ποιες είναι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα μάλλον της δράσεώς μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλησα να δώσω μερικά παραδείγματα. Οι δράσεις μας για την προστασία της επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τον ΙΦΑΟ Έχουμε διεθνή προγράμματα για την εξάλληψη ε, ε, ζωονόσων, για παράδειγμα την πανόλη των βοηδών που είχε χτυπήσει και την Ευρώπη τον περασμένο αιώνα με ε, πολύ βαρύ τρόπο. Προχωρούμε και για την εξάλληψη του αυτόδος πυρετού, με, επίσης για την εξάλληψη της λύσας στα σκυλιά και με τον ΦΑΟ για την εξάλληψη της πανόλους των μικρών μυρικαστικών. Εργαζόμεθα επίσης για την αντιμετώπιση των βιολογικών ε, κινδύνων που προέρχονται είτε από ατυχήματα είτε από τρομοκρατικές επιθέσεις. Τον Ιούνιο στο Παρίσι διεξήχθη διεθνής διάσκεψη με συμμετοχή ε, των κτηνιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δημόσιας υγείας αλλά και με ε, διοκτικές αρχές, με αρχές που αντιμετώπιση τρομοκρατία κτλ. Για να αντιμετωπιστούν τέτοια θέματα απειλών. Έχουμε επίσης πρόγραμμα μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα για την αντιμετώπιση του Παστοράδη, ιδίω στο Σαχέλ, διότι ο Λαό του Σαχέλ είναι εύκολα θύματα στρατολόγηση από εξτρεμιστές και οι δράσεις μας είναι ουσιώδεις για την πρόληψη της τρομοκρατίας και για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιούνται οι ευκαιρίες αυτές από εγκληματίες. Προτείνουμε τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεις για την πρόληψη των κρίσεων που οφείλονται στον ιό έμπολα, κάνοντας χαρτογράφηση της παρουσίας του ιού στην Αφρική και σε φορείς, άγριους φορείς δηλαδή, αλλά και με εμβολιασμό των, ε, κινδύνων, των ε, πληθυσμών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο. Διευκολύνουμε και το εμπόριο. Με την ύπαρξη των κανόνων μας που εφαρμόζονται καταρχήν από όλες τις χώρες μέλη μας, η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση, όντας μία από τις περιφέρειες του κόσμου που εφαρμόζουν περισσότερο, συμμορφώνονται περισσότερο με τους κανόνες του οργανισμού μας και λόγω του περιεχομένου των κανόνων αυτών δεν κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ε, προσφυγές ε, στο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τα εγγραφεία που έχουμε στη Μόσχα, στο Καζακστάν, στις Βρυξέλλες, στον Παμακό, στην Τίνιδα και στον Αερόμπι είναι σημαντικά σημεία ενίσχυσης των προγραμμάτων που όλα τα προγράμματα αυτά ωφελούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και από τους μεγαλύτερους δωρητές του οργανισμού μας μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας με ε, επιστημονική συνεργασία, με σεμινάρια και ενημέρωση ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου επίσης μας βοηθεί να συνδέουμε τις ε, άλλες χώρες στις ψηφοφορίες και επίσης εξασφαλίζει την παρουσία εκπροσώπων τους σε όλες τις συζητήσεις μας και στις γενικές συνελεύσεις μας, κάτι πολύ σημαντικό για να συνδεθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες με την δημιουργία των, με την θέσπιση των ίδιων των κανόνων και τέλος συνεργαζόμαστε και με την Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας για την αντιμετώπιση ε, ζωνώσεων και στην Ασία και στην Αφρική και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι το Ευρωκοινοβούλιο ε, ενέκρινε 3,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεων για την ε, καλή διαχείριση της αντιμετώπισης των ζωνώσεων στην Αφρική και για προγράμματα προλήψεως της εξάπλωσης της λύσας. Και βεβαίως αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι παρά μια αρχή. Άρα ας συνεργαστούμε με τρόπο αμοιβαίως επωφελή, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλή διαχείριση, την καλή τη χρηστή διοίκηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα έχουμε ελεγχθεί πρόσφατα από γραφείο ορκωτών λογιστών πάρα πολύ αυστηρό και αυτοί ήλεγξαν τους έξι πυλώνες και μας ε, και ενέκριναν, μάλλον ε, μας ε, έδωσαν κάθε βαθμολογία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Βαλά. Φυσικά η ευημερία των ζώων, η υγεία των ζώων είναι το μίσο στους οποίους ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει αξιοσημείωτα επιτεύγματα και γι' αυτό και ο δικός σας οργανισμός έχει μεγάλη σημασία. Πέντε συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, έξι. Ένα λεπτό καθένα παρακαλώ. Ο κύριος Βοητσεχόφσκι, αλλά θερμά σας παρακαλώ ένα λεπτό μόνο. Ευχαριστώ. Τι να πρώτο προλάβουμε σε ένα λεπτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του Γενικού Διευθυντού. Λακωνικότατα πάντως. Μιλήσατε για τις δυσκολίες ε, εφαρμογής των διατάξεων για την ευημερία των ζώων. Ιδιαίτερα στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες. Νομίζω ότι πιο ισχυρό επιχείρημα είναι ότι η κακομεταχείριση των ζώων στην κτηνοτροφία, στη μεταφορά, αλλά και κατά τη διάρκεια της φαγής, προκαλεί κίνδυνο και στην υγεία των ανθρώπων, γιατί το στρες, το άγχος ε, που βιώνουν τα ζώα σε περίπτωση κακομεταχείριση μετατρέπεται σε τοξίνες ε, και σε ένα κρέος ε, που είναι επικίνδυνο και για τη δημόσια υγεία. Οπότε, αν δεν αρκεί το ανθρωπιστικό επιχείρημα για την ευημερία των ζώων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το επιχείρημα της υγείας, της ανθρώπινης υγείας. Ελπίζω να μην προσβληθούν οι Ρουμάνοι συνάδελφοι με αυτό που θα πω, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ρουμανία και φαίνεται από τις επιστολές ε, που στέλνουν από τη Ρουμανία οργανώσεις προστασίας των ζώων και υπάρχει τεράστιος αριθμός αδέσποτων σκυλιών στην ε, Ρουμανία και φυσικά μερικά θανατώνονται αλλά υπάρχει τεράστιος αριθμός και μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχει σύστημα ταυτοποίησης ε, και πολύ σωστά αυτών των αδέσποτων σκυλιών. Ε, βέβαια, πολύ πολλά θετικά εγκαταλείπουν τα σκυλιά γιατί δεν μπορούν να αναλάβουν το κόστος ε, συντήρησής τους. Ε, αλλά έτσι πολλά διαφεύγουν και από τους ελέγχους, από τους εμβολιασμού, κάτι που δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία. Και από τη Ρουμανία ειδικά έχουμε πολλές επιστολές ε, που μας επισημαίνουν αυτό το πρόβλημα. Έχετε γνώση της κατάστασης και ποια είναι η προσέγγιση του οργανισμού σας προς το θέμα αυτό. Ναι, ξέρω ότι ασχολείστε ιδιαίτερα αυτό το θέμα και θα μπορούσατε να αναπτύξετε για πολλή ώρα αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Η ε, κυρία Αγγιλέρα, ένα λεπτό παρακαλώ κι εσείς. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και το Γενικό Διευθυντή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπατε, ότι εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαστε με τα θέματα της ευημερίας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό επηρεάζει άμεσα τους κτηνοτρόφους μας. Και ακριβώς ε, με τις εισαγωγές και τη μη τήρηση αντίστοιχων προδιαγραφών στις τρίτες χώρες είχαμε αθέμητο ανταγωνισμό. Θεωρείτε ότι έχει μειωθεί αυτή η κατάσταση και ότι έχει αυξηθεί αυτή η ανταγωνιστικότητά μας γιατί στις διμερείς συμφωνίες οπότε λαμβάνει υπόψη το θέμα της ευημερίας των ζώων. Οπότε θεωρώ ότι εξακολουθεί να υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό και διαφορά στην ανταγωνιστικότητα ει βάρο των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων. Επίση, ε, αναφερθήκατε σε μια παγκόσμια στρατηγική για την ευημερία των ζώων. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα στοιχεία. Και πώ θα συνδυαστεί με την ευρωπαϊκή στρατηγική τη ευημερία των ζώων για την επόμενη τριετία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ. Η παρουσίασή σας ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την ε, Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Γιατί εδώ και μια διετία αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι οξύ ιδιαίτερα στις βαλτικές χώρες και την Πολωνία. Οι βαλτικές χώρες υποφέρουν ε, από αυτή την επιζώτια, την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων που δυστυχώς ε, εξαπλώνεται και δεν περιορίζεται. Τι θα μπορούσατε να μας προτείνετε, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, ένα πρόβλημα ιδιαίτερα οξύ στις Βαλτικές χώρες και την Πολωνία. Άκουσα ότι έχει προκηρυχθεί ε, διαγωνισμός για την ε, Παρασκευή εμβολίου για την ζώνη αυτή. Είναι προτεραιότητα όμως η καταπολέμησή της. Ποια είναι η δική σας γνώμη και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και στα άγρια γουρούνα και στα άγρια γουρούνα, στους αγριόχειρους. Είναι σωστή αυτή η προοπτική και η προσέγγιση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα που έχει το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο κατά κεφάλι ε, σε συνδυασμό με τον πληθυσμό από στον κόσμο, τις κάτω χώρες. Και μάλιστα η μεταφορά αυτών των ζώων ε, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά ζωντανά ζώα. Οπότε μας ενδιαφέρει το θέμα της ευημερίας των ζώων, το θέμα της μικροβιακής αντοχής, αλλά και τα κρούσματα νέων ε, ζώων όσων, VSR, SPL. Επίσης, στην τρίτη παγκόσμια διάσκεψη για την υγεία των ζώων και την ευημερία των ζώων, που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων στην Κουάλα Λουμπούρ, προέκυψε η σύσταση να, γίνει, να οργανωθεί με παγκόσμια στρατηγική για την ευημερία των ζώων και την υγεία των ζώων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν έχει προτείνει ακόμη νέα στρατηγική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, στην παρουσίαση Ακούσαμε ότι ο μιλητής ήταν υπέρ εμβολιασμού ε, για τον αυθόδη πυρετό ε, των χείρων αντί να σκοτώνται τα ζώα. Το 2001 και 2005 μάλλον είχαμε, 2001 είχαμε αυτή την επιζωτία. Λοιπόν, την εκριζώσαμε την ασθένεια και γι' αυτό μπορέσαμε να εξάγουμε το κρέας. Αν είχαμε εμβολιάσει θα θεωρούσαμε ότι θα ήμασταν φορείς ασθένειας και θα μπορούσαμε να εξάγουμε το κρέας. Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο λοιπόν για τη μη διεξαγωγή εμβολιασμών. Ε, μπορείτε να σχολιάσετε. Θα πάω και εγώ στη Ρουμανία. Υπάρχουν πολλοί αδέσποτοι σκύλοι και 22% πάσχουν απολύσει από ό,τι λέγεται. Ποια είναι η άποψή σα, τι, τι πρέπει να γίνει. Λόγω της ελεύθερης διακινήσεως των ανθρώπων και επειδή η λύσα είναι ζωονόσος, σημαίνει ότι μπορεί να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να γίνουν βήματα και προτείνω όλα αυτά τα σχολιά να ε, εξουδετερωθούν, να εξοντωθούν. Ο κύριος Δαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Βαλά, όχι μόνο για την ομιλία του, αλλά κυρίως για τη δράση του. Γιατί η πολύχρονη πείρα του στη, στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και η κορυφαία του θέση έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε αυτόν τον οργανισμό. Ε, οπότε, αν μη τι άλλο, θερμά ευχαριστώ για την προσφορά σας, ε, ενώ θα μπορούσατε να έχετε μια πολύ πιο ήρεμη ζωή. Πιστεύετε ότι οι κλιματικές αλλαγές ε, αυξάνει τους υγειονομικούς κινδύνους ε, για το ευρωπαϊκό ζωικό κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και εσάς κύριε Γενική Διευθύντα. Και λυπούμε διότι σε ένα μέρος της παρουσιάσεως σας ήμουν πούσα σε άλλη επιτροπή. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος των κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η πραγματικότητα σε πολλές χώρες μέλη είναι ότι όλο και, λιγότερο, και λιγότεροι κτηνίατροι ε, ασχολούνται με τα μεγάλα ζώα παραγωγής, ιδίως βεβαίως ε, στο Ενωμένο Βασίλειο αλλά και σε πολλές άλλες χώρες μέλη. Και ποια θα είναι η επίπτωση στην ε, υγεία και στην ευημερία των ζώων. Δεύτερο, η διαθεσιμότητα φαρμάκων και εμβολίων ποιες δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε στο επίπεδο των πολιτικών για να υπάρχει ε, διαθέσιμη αρκετή ποσότητα ε, ιατρών. Τώρα, ο ιός Σμάλενμπεργκ, πού βρίσκεται η κατάσταση, διότι υπάρχει κενό στην επιστήμη, εμφανίστηκε στην Ιρλανδία και μετά εξαφανίστηκε και κανείς δεν κατάλαβε πώς και γιατί. Από την άλλη μεριά, η ε, ζωονόσους γιούνες και η σχέση της με την ανθρώπινη υγεία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ. Ε, έχουμε στους ζωικούς πληθυσμούς σημαντικές αλλαγές. Μερικοί μειώνονται, άλλοι αυξάνονται κάτι που μπορεί να δημιουργήσει απειλές για βιολογική, στη βιολογική ισορροπία. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της ευημερία των ζώων ή ε, η έλλειψη ευημερία ε, ως απειλή στην ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, συνθήκες ε, μεταφοράς των ζώων ή σφαγής. Το κρέας των ζώων μπορεί να υποστεί αλλαγές και αλλοιώσεις εξαιτίας ε, κακής μεταφοράς με αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτού του κρέατος να δημιουργήσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Μπορούμε όμως να μειώσουμε αυτό τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία με κατάλληλους ελέγχους και επιθεωρήσεις των προϊόντων αυτών, του κρέατος δηλαδή. Και τα κείμενα και οι διατάξεις εκτινετρικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπουν αυστηρότατους ελέγχους για προϊόντα που προορίζονται στην ανθρώπινη κατανάλωση. Και αυτοί οι έλεγχοι και επιθεωρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν αυτούς τους κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία. Δυστυχώς όμως Δυστυχώ όμως το γεγονός ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δεν αναγνωρίζει τι εμπορικές συμφωνίες τι διατάξει για τις ευημερίε των ζώων, με εξαίρεση τι τελευταίε εξελίξεις που σας ανέφερα, δεν μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε εμπορικές διαφορές σε περίπτωση καταπάτησης των διατάξεων Τη ευημερία των ζώων. Οπότε η στρατηγική μα είναι να αποφασίσουμε τους πολιτικούς ηθήνοντε όταν διαπραγματεύονται διμερεί συμφωνίε να συμπεριλάβουν και την ευημερία των ζώων σε αυτές τις διμερείς συμφωνίε. Για να διευκολύνουν την εφαρμογή των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων στις διμερείς συμφωνίες. Αυτό είναι το καλύτερο όπλο που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο επιχείρημα. Είναι η επίδραση του πληθυσμού των τρίτων χωρών στις κυβερνήσεις. Και εκεί έχουμε θεαματικές εξέλιξεις. Για παράδειγμα, στην Κίνα, σε μια χώρα δηλαδή που δεν υπήρχαν διατάξεις πριν από 10 χρόνια για την ευημερία των ζώων, σήμερα η Κίνα υιοθετεί όλο και πιο αυστηρά μέτρα για την ευημερία των ζώων. Και δεν είναι η μόνη αναδυόμενη οικονομία που θεσπίζει τέτοια μέτρα. Υπάρχει λοιπόν μια παγκόσμια εξέλιξη και μια πολύ θετική και ενθαρρυντική τάση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο δικό μας οργανισμό και στον συστηματικό διάλογο που έχουμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με την ευημερία των ζώων. Και μιλώ για μετριοπαθείς οργανώσεις, όχι τις εξτρεμιστικές. Έχουμε λοιπόν μόνιμους δεσμούς με τις οργανώσεις αυτές και με συνεργασία μαζί τους προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποια πρόοδο. Και κάτι τέτοιο γίνεται προς όφελος και των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις πιο δεσμευτικές παγκοσμίω διατάξεις για την ευημερία των ζώνων. Σε ό,τι αφορά τα δέσποτα, τα λανιάρικα σκυλιά. Σε πολλές βαλκανικές χώρες μας βοηθά η Γενική Διεύθυνση Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να οργανώσουμε σεμινάρια και επιμόρφωση στις Βαλκανικές χώρες. Και μάλιστα οι εθνικοί φορείς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτά τα σεμινάρια, για τον έλεγχο των αδέσποτων σκυλιών. Και μάλιστα στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων έχουμε ολόκληρο κεφάλαιο για το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων σκυλιών. Προκειμένου να αποφύγουμε την εξάπλωση της λύσας για να μην συνεχίζεται η εξάπλωση της λύσας εξαιτία των αδέσποτων σκυλιών. Σε μερικές περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας κανόνες και πρότυπα που μας επιτρέπουν κάποιες αξιοπρεπείς δράσεις, οι κυβερνήσεις μπορούν να αποφασίσουν εξολόθρευση των ζώων, θανάτωση των ζώων υπό όρους, κυρίως λόγω κινδύνου της λύσας. Και αυτό επιτρέπεται και είναι δυνατό με σεβασμό των παγκόσμιων κανόνων. Βέβαια, καλό θα ήταν να δώσουμε έμφαση στην διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, επιμένοντα σε παράγοντε που, που περιορίζουν την αναπαραγωγή του για να μην χρειαστεί να κατεφύγουμε αργότερα στη θανάτωση. Αυτό και είναι σημαντική η διοργάνωση σεμιναρίων και κατάρτιση. Και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μα βοηθά στην οργάνωση αυτών των σεμιναρίων των επιμορφωτικών, κυρίω στι Βαλκανικέ χώρε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση μιας παγκόσμιας στρατηγικής για την ευημερία των ζώων, όντως στην παγκόσμια διάσκεψη που έγινε στην Κουάλα Λουμπούρ υιοθετήθηκε μια σύσταση υπέρ της ε, θέσπισης μιας τέτοιας στρατηγικής. Γι' αυτό και το ανέφερα προηγουμένως. Και μάλιστα θα έχουμε και παγκόσμια διάσκεψη ε, για την ευημερία των ζώων στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού το Δεκέμβρη του 2016. Εκεί θα προτείνουμε στις χώρες που συμμετέχουν στη διάσκεψη την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής, της παγκόσμιας στρατηγικής για την ευημερία των ζώων και φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχει στις προκατακτικές συζητήσεις. Σε ό,τι αφορά την πανόλη των χείρων, την αφρικανική πανόλη των χείρων, δυστυχώς δεν υπάρχει εμβόλιο για τη ζώνος αυτή αφενός και αφετέρου πρόκειται για μία νόσο που ε, συνδέεται και με τα αγρία Οι αγριόχειροι, για παράδειγμα, συμβάλλουν ιδιαίτερα στην εξάπλωση του, της πανόλης ε, των χείρων. Μάλιστα, η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων χτύπησε την Ισπανία και την Πορτογαλία πριν από μία εικοσαετία. Και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν εμβόλια και παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλος πληθυσμός αγριοχείρων, τελικά η Ισπανία και η Πορτογαλία κατάφεραν να απαλλαχθούν από την ζώνη αυτή και εδώ και 20 χρόνια δεν έχουν ε, κρούσματα ε, τέτοιες αφρικανικές πανόλης χείρων και έτσι μπορούν να εξάγουν το υπέροχό τους ζαμπόν στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Τι μπορούμε να προτείνουμε. Διαχείριση του πληθυσμού των αγριοχείρων με σωστό και κατάλληλο τρόπο. Δηλαδή η μαζική θανάτωση αγριοχείρων ε, οδηγεί στο στην μετάδοση σε άλλες ζώνες, σε περίπτωση που ξεφύγουν μερικοί αγριόχειροι από τη σφαγή. Βέβαια, η μη διαχείριση του πληθυσμού των αγριοχείρων ε, ευνοεί την εξάπλωση της νόσου, γιατί όταν είναι πολύ αγριόχειροι η μόλυνση είναι πολύ πιο συχνή. Θα πρέπει να έχουμε συμφωνίες λοιπόν και με τους κυνηγούς. Και τον Ιούνιο οργανώσαμε ένα σεμινάριο με τις ευρωπαϊκές χώρες και εκπροσώπους των κυνηγών και εθνικές ομοσπονδίες κυνηγών και κυνηγητικούς ομίλους και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ τους. Και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι σε μερικέ χώρε κυνηγητικοί σύλλογοι δεν είχαν καμία επαφή με κτηνιατρικέ υπηρεσίε. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή την συνεργασία για να επιμορφώσουμε του κυνηγού ώστε να εντοπίζουν αυτή την όσο και φυσικά να επενδύσουμε και στην έρευνα για να βρούμε εμβόλιο για, τον αυθόδη, πυρετό, για την αυθόδη των χείρων. Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι πολύ δαπανηρό. Και φυσικά, στα χειροστάσια θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλοι έλεγχοι ασφάλειας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τους όρους της βιοασφάλειας ή να υποχρεώνουν τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους τους να τους εφαρμόζουν, παρόλο που είναι δαπανηρή εφαρμογή αυτών των όρων βιοασφάλειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των νέων όσων και των κλιματικών αλλαγών, το γεγονός ότι οι χειμώνες είναι πιο θερμοί επιτρέπει στους φορείς, τα μεγάκια, τα κουνούπια, να επιβιώνουν το χειμώνα. Ενώ στο παρελθόν που είχαμε πιο κρύους χειμώνες δεν επιβίωναν οι φορείς. Από τη στιγμή που επιβιώνουν όμως τα έντομα οι φορείς, επιβιώνουν και τα μικρόβια, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο της μετάδοσης των ασθενειών. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε πιο θερμούς, πιο ήπιους χειμώνες. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν την εξάπλωση των νόσων. Αλλά φυσικά το θέμα αυτό επιδέχεται πολύ ωραία συζήτηση. Επίσης, ε, οι κτηνίατροι δεν πηγαίνουν σε απομονωμένες ζώνες. Δεν υπάρχουν αρκετοί κτηνίατροι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα τις ορεινές περιοχές, τις πολύ ψυχρές περιοχές. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν μέτρα και να ενθαρρύνουν τους ε, κτηνιάτρους να εγκαθίστανται και σε απόμακρες περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό για την υγεία όλων μας. Και υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι. Μερικές ε, χώρες πληρώνουν τους κτηνιάτρους με δημόσια κονδύλια και βρίσκουν υποψηφίους και για τις ε, απομακρυσμένες περιοχές. Τώρα, για τα άγρια ζώα, άγρια πανίδα, σε μερικές περιπτώσεις ε, όντως θα πρέπει να την περιορίσουμε την άγρια πανίδα. Σε άλλες περιπτώσεις όμως θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Δεν είναι η ίδια η ρυθμή ανάπτυξη ε, των διαφόρων πληθυσμών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή διαχείριση, ε, περιβαλλοντική, αλλά και συμφωνίες με τις κυνηγετικές οργανώσεις, γιατί όταν έχουμε υπερβολική αύξηση των άγρων πληθυσμών, οι κυνηγοί θα μας βοηθήσουν να τους ελέγξουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Υγεία των Ζώων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτόν τον οργανισμό γιατί η συμβολή του είναι τεράστια σε θέματα υγείας των ζώων. Το είπε προηγουμένως και ο κύριος Ντάντα. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο οργανισμός σας. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο αγαπητοί συνάδελφοι. Απαλλαγή, απαλλαγή για τον προπολογισμό του 2014. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση του κυρίου Σανή. Πολύ σημαντική γνωμοδότηση, γιατί μερικές φορές δεν υπάρχει συνεννόηση, κατανόηση ε, για, ως προς την αναγνώριση που θα πρέπει να δοθεί στη Γεωργία και το σημαντικό ρόλο της. Υπάρχει μερικές φορές διαφορετική αντίληψη και ερμηνεία για το θέμα αυτό. Θα δώσω το λόγο στο συντάκτη της γνωμοδότησή μας, τον κύριο Σανί, τον οποίο θέλω να παρακαλώ να είναι σχετικά σύντομος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σωστά τα είπατε. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και ότι μέσω του Κοινοβουλίου όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση που κρατεί στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Να σας ενημερώσω. Το έργο στον αφορά την απαλλαγή στον τομέα της Γεωργίας συνεχίστηκε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις συστάσεις τους. κυρία Κουτάρ που είναι πίσω μου. Βασικά, άγγελος ήταν. Βοηθός. Μετά την πρώτη μας συζήτηση, λάβαμε την έκθεση του λεκτικού συνεδρίου. Έτσι αποκτήσαμε και μια άλλη άποψη για τις επιδόσεις. Θα αναφερθώ στα διάφορα σημεία. Θα θέσω κάποια ερωτήματα. σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που έχετε όλοι σε όλες τις γλώσσες. Πρώτα απ' όλα, παράγραφος 6. Την πολλαπλή συμμόρφωση. Μήπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας απαντήσει στο δίλημα που αναφέρεται. Σφάλματα όσον αφορά την συμμόρφωση. Έγκαιρη δήλωση μετακινήσεως ζώων. Τήρηση προθεσμιών. Αυτά τα σφάλματα δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα, συμφωνώ. Τι ούτω τρόπος αν μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων όσον αφορά, αν αφαιρέσουμε το ποσοστό σφαλμάτων από την πολλαπλή συμμόρφωση, από το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης, ε, πάμε στο 1,2% για τα EGF και 6% για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Άρα έχουμε βελτίωση. Εν συγκρίση με πέρσι. Το πρώτο σημείο ήταν αυτό. Το δεύτερο αφορά την παράγραφο 10. Το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσε να εξηγήσει την προσέγγιση όσον αφορά τις επιδόσεις που ακολούθησε για τις δαπάνες για τη Γεωργία. Παράγραφος 13. Ζητά από τα κράτη-μέλη να ε, απλουστεύσουν την κατάσταση αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι ένα από τα βασικά εμπόδια για τις επενδύσεις στην Ήπεθρο. Τα κράτη-μέλη λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μειώσουν βασικά τον περίπλοκο χαρακτήρα των μηχανισμών, δηλαδή να επιφέρουν απλούστευση, κάτι που ζητούμε και στην παράγραφο 14, μετά παράγραφος 16. Η σημασία συγκρίσιμων δικτών επιδόσεων και στόχων όσον αφορά τις επιδόσεις. Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις στο Συμβούλιο δεν θέλουν να κινηθούν τίτο τρόπο σε διαφόρους τομείς. Σίγουρα δεν, με, δεν μπορούν να προσμετρηθούν οι επιδόσεις αν δεν είναι συγκρίσιμες. Παρατήρηση παριθμών 5. Παράγραφος 23. Ζητούμε επικαιροποίηση όσον αφορά βελτιώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση. Έκτο σημείο. σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας πει αν είναι πιο πλήρες οι πληροφορίες για το ΕΠΑΡΤ και για τα στοιχεία για τη 2014. Όταν κατατίστηκε αυτό το, αυτή η ενημέρωση ήταν επικαιροποιημένα τα στοιχεία. Αυτό το αναφέρουμε στην παράγραφο 24. Τέλος. Έλλειψη συνοχής. Μεταξύ ετησίων και πολυετών προσεγγίσεων στην παράγραφο 25. Το λεκτικό συνέδριο καλείται να μας ενημερώσει πώς θα, θα αναπτύξει μια μεθοδολογία πολιετούς αναλύσεως. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά θέματα που ήθελα να θίξω σε αυτό το στάδιο και θα ήθελα να ακούσω σχόλια και παρατηρήσεις από τους συναδέλφους και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Ήδη συζητήσαμε το θέμα και παλιά. Λοιπόν, παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Κυρία Γκαρσία έχει το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Βαρκάλ ως αντιπρόεδρος έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είναι στο Λουξεμβούργο σε μια συνάντηση της ΚΟΣΑΚ και ήθελε λοιπόν να τον αντικαταστήσω σήμερα σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα του προπολογισμού. Ήθελε καταρχάς να πω στον κύριο Τσάνι ότι εκτιμά τα μάλα το επιτελεστέν έργων και θεωρεί ότι σωστά τονίζει τον κοινωνικό αντίκτυπο της ΚΑΠ και τον αντίκτυπο που έχει στην Ήπεθρο και θέλει να τονιστεί και μείωση των σφαλμάτων από το 2013 στο 2014 κυρίως διότι το 2014 έχουμε μεταβατικό έτος γιατί είχαμε την περίοδο 2000, ε, πάμε στην επόμενη περίοδο πληρωμών από 2015 μέχρι 2020 και αυτό είναι σημαντικό. Συμφωνεί λοιπόν με τα σχόλια της εκθέσεως για τη δυσκολία δρομολογήσεως πολιετών προγραμμάτων με μια αξιολόγηση ετήσια που γίνεται των πολιετών δημοσιονομικών πλαισίων και χρειάζεται απλούστευση των συστημάτων διαχείρισης. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διατυπώσεις για τις άμεσες πληρωμές. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Επιτρόπου Χόγκαν και τη δήλωση ότι θα γίνουν πολλές απλουστεύσεις, επιτέλους κάποτε πρέπει να πραγματοποιηθούν. Επίσης είπαμε θα αυξηθούν οι επιτόποι έλεγχοι το 2017, παρόλο που το ποσοστό σφάλματο είναι κάτω από το 2%. Ο κύριος Βαλκάρσελ θεωρεί ότι η απλοποίηση τη κοινή πολιτική πολιτικής και φυσικά θα εξετάσει πιο ενδελεχώς το κείμενο στο μέλλον. Ε, μπορεί να υποβάλει και κάποια τροπολογία για την απλούστευση των διοικητικών ελέγχων ή την περιπλοκότητα που έχει το θέμα του πρασινίσματος γεωργίας και κυρίως το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτός στους μελλοντικούς ελέγχους. Σας ευχαριστώ κύριε Σελιμόβιτς. Ευχαριστώ για την πρότασή σας. Εμείς θεωρούμε ότι τα βασικά στοιχεία της προτάσεως είναι θετικά και συμφωνούμε. Βέβαια έχουμε και ορισμένα σημεία όπου θεωρούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε ακριβή αποτελέσματα ελέγχου των απατών και ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. Διότι είμαστε Επιτροπή Γεωργίας και βεβαίω η Επιτροπή Γεωργίας δαπανά χρήματα, αλλά η ιδέα ότι τα χρήματα αυτά σπαταλώνται πρέπει να, πρέπει να ε, αντιστραφεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καταθέτουμε ορισμένες τροπολογίες που ναι μεν δεν τροποποιούν τη βασική γραμμή της πρότασης, ωστόσο ε, επιτρέπουν ακριβέστερες διατυπώσεις. Σας ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει ολόκληρο επιτελείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Το εκτιμούμε ιδιαίτερος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δίνετε το παρόν και παρακολουθείτε τις ε, συζητήσει που γίνονται στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλωσορίζουμε το σχέδιο εκθέσεω του εισηγητού. Καλύπτει, πιστεύω, τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο το παρόν της απαλλαγής να αναφερθώ σύντομα στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Κατά την άποψή μας, γενικά, είναι ενθαρρυντική και για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μειωτική τάση όσον αφορά τα σφάλματα και τους δύο πυλώνες, τον πρώτο και τον δεύτερο. Επίσης σημειώνουμε ότι το συνέδριο έκρινε γενικά θετικά τη διαχείριση τη κοινή αγροτική πολιτική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλαβε υπόψη τη βελτίωση που πετύχαμε μαζί με τα κράτη-μέλη. Τα συστήματα διαχείριση και ελέγχου, ε, το ολοκληρωμένο σύστημα για τι πληρωμέ να, να βελτιωθεί. Ο εισηγητή αναφέρθηκε σε κάποια θέματα. Έχω κάποια σχόλια σχετικά. Την πολλαπλή συμμόρφωση πρώτα απ' όλα. Πράγματι, λάβατε εσεί απόφαση στα πλαίσια τη μεταρρυθμίσεω τη ΚΑΠ ότι τώρα στον οριζόντιο κανονισμό αναφέρεται ότι πολλαπλή συμμόρφωση, τα σφάλματα της πολλαπλής συμμορφώσεως δεν λαμβάνονται υπόψη σαν προβλήματα επιλεξιμότητας. Συνεπώς δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό σφαλμάτων. Το Λεκτικό συνέδριο ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση. Ανακοίνωσε ότι από το 2015 το οικονομικό έτος και πέρα το 2015 συμπεριλαμβάνει την πολλαπλή συμμόρφωση θα συναφή ζητήματα τα ποσοστά σφαλμάτων. Το είχαμε προβλέψει αυτό κάπως. Θα είχαμε λοιπόν για τον πρώτο πυλώνα το 2014 2,2% να ακολουθούσαμε την προσέγγιση του ελεκτικού συνεδρίου, τη νέα. Οπότε πλησιάζει και στο όριο του 2% εφαρμογής, που είναι η ιερή αγελάδα του εγχειρήματο. Για τον πρώτο πυλώνα το 2014 τα πράγματα εξελίχθησαν αρκετά θετικά. Παρόμοια τάση έχουμε για το δεύτερο πυλώνα. Χωρίς πολλαπλή συμμόρφωση, όπως είπε ο εισηγητή, το ποσοστό σφαλμάτων είναι 6%, πολύ υψηλό, αλλά αρκετά πιο χαμηλό από ό,τι ήταν τα προηγούμενα έτη, όταν πριν από δύο χρόνια είχαμε 7,9% φερρυπίν. Και εκεί νομίζω ότι σωστά πηγαίνουν τα πράγματα, από σωστή κατεύθυνση. Για την απλούστευση και την ανάπτυξη υπαίθρου, σας διαβεβαιώνω ότι ο Επίτροπος Χόγκαν είναι αποφασισμένος να επεξεργαστεί το θέμα. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Γενική Διεύθυνση για τα θέματα γεωργίας ολοκληρώνει διαδικασία εγκρίσεων για τα 118 προγράμματα αναπτύξεως της υπαίθρου που θα πρέπει να υλοποιηθούν και ότι οι δραστηριότητες απλουστεύσεως θα εφαρμοστούν από τη στιγμή που θα λήξουν αυτά. Τα τελευταία προγράμματα έχουν ήδη δρομολογηθεί, πιθανότατα μέχρι το τέλος του ενεστώτος έτους ε, όλα τα προγράμματα θα εγκριθούν. Ταυτόχρονα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ομάδα εμπειρογνωμάνων ψηλού επίπεδου υπό τον κύριο Σιμ Κάλλας, πρώην Επίτροπο και Αντιπρόεδρο, για να εξετάσουν την πιθανότητα απλουστεύσεως όχι μόνο της αναπτύξης υπαίθρου, αλλά όλων των διαθροτικών ταμείων της Ευρώπης και των επενδυτικών ταμείων. Και είμαι πεπισμένος ότι θα δούμε τα αποτελέσματα του έργου αυτού κατά τη διάρκεια του 2016. Ο συγκεκριτής είπε ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων μας και των μέτρων μας και η υποβολή αναφορών για τις επιδόσεις μπορεί να γίνεται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν συγκρίσιμες προδιαγραφές. Επ' αυτού Βάσει αποφάσεως που λάβατε ως συνομοθέτης στα πλαίσια της μεταρρυθμίσεως, στην ΚΑΠ έχουμε ετοιμάσει κοινό πλαίσιο παρακολουθήσεως και εξολογήσεως με κοινά αποτελέσματα και δείκτες συνεπιών που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή τη φορά θα έχουμε πολύ πιο στέρεη βάση για την μέτρηση επιδόσεων στην ΚΑΠ. Ο εισηγητής έθεσε ένα ερώτημα όσον αφορά το ΙΠΑΡΤ και είμαι εσύ λυπούμε που δεν μπορώ να σας δώσω τώρα λεπτομέρειες σε αυτή τη συνεδρίαση αλλά θα διαβιβάσω τα σημεία αυτά και θα δώσω απαντήσεις διμερώς στον εισηγητή ούτω ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες στα πλαίσια της όλης προσπαθίας που καταβάλλεται, του όλου εγχειρήματο. Να πω τέλος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τις απόψεις του εισηγητού που εκφράζονται στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως ότι προσμέτρηση των επιδόσεων κυρίως σε μια πολιτική για την ΚΑΠ ετησίως είναι κάτι μη ρεαλιστικό στόχος. Οι επενδύσεις που γίνονται όσον αφορά τη στήριξη εισοδήματος και για διαφορετική υποστήριξη την ανάπτυξη της υπαίθρου δίνουν καρπούς όχι εντός μερικών εβδομάδων και μηνών, αλλά μετά από σειρά ετών και καμιά φορά μετά από δεκαετίες. Γι' αυτό στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ξεκινήσαμε να αναφέρουμε τις επιδόσεις της ΚΑΠ σύμφωνα με πιο μακροπρόθεσμη προπτική. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε πιο αξιόπιστη και ρεαλιστική εικόνα των επιτεγμάτων της ΚΑΠ και των ελλείψεων αυτής και που χρειάζονται βελτιώσεις. Λοιπόν, για να τα πω όλα μαζί, αν κατακλείδει το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που υπευλήθη κατά την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αποτελεί πολύ στέρη βάση για μια ρεαλιστική αξιολόγηση των προσπαθειών για την υλοποίηση της ΚΑΠ και των δαπανών για αυτό το σκοπό που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν το 2014, εξακολουθούμε να είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε με οδήποτε τρόπο, αν αυτό παραστεί αναγκαίο και το ζητήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ο συντάκτης γραμματότησης μας τώρα, κύριο Σάνι. Χρόνο φίδου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τους ε, συναδέλφους για τα ευγενικά τους λόγια. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά πράγματα σε αυτά που είπα προηγουμένως. Υπό το φως ε, και των ε, τελευταίων παρεμβάσεων που ακούσαμε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να νιώθει υπερήφανη για την κοινή γεωρική πολιτική της και την εξέλιξη αυτής της τελευταίες δύο δεκαετίες. Και το λέω παρά τις αντιρρήσεις που ακούσαμε και τις διαφωνίες είναι μεγάλο το επίτευγμα της ΚΑΠ και έχει διαμορφώσει μια διαφορετική Ευρώπη από αυτή που υπήρχε πριν την θέσπιση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Και η κοινή γεωργική πολιτική είναι όχι μόνο η παλαιότερη αλλά και πιο εκλεπτισμένη κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις μας. Προς αυτή την κατεύθυνση επικεντρωνόμαστε και αυτό προσπαθούμε. Και οι τάσεις είναι γενικώ ενθαρρυντικές. Συμφωνώ με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το σχέδιο της γνωμοδότησης που υπέβαλα είναι απλώς η βάση για τη συζήτηση. Και προσκαλώ τους συναδέλφους να το λάβουν υπόψη. Και ναι κύριε Σιλιμόβιτς και εσείς και όλοι οι συνάδελφοι παρακαλώ υποβάλλετε τις προτάσεις σας. Δεν θέλω να διστάσετε καθόλου γι' αυτό. Και δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ. Έχουμε και το σχέδιο έκθεσης. Δεν ανέφερα ούτε κουβέντα γι' αυτό. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα αλλά θα πρέπει ε, το σχέδιο έκθεση να το δούμε από κοινού με τις συζητήσει που γίνονται και τις παρατηρήσεις που υποβάλλεται. Πιστεύω ότι αν επικεντρωθούμε σε τρεις βασικούς άξονες, σε τρία βασικά σημεία, θα είμαστε στο σωστό δρόμο. Δηλαδή, πρώτον, πώς θα ελέγξουμε τις δαπάνες, γιατί είναι καθήκον μας απέναντι στους φορολογουμένους. Θα πρέπει τα κοινοτικά κονδύλια να πιάνουν τόπο, να γίνεται χρηστή διαχείρισή τους. Και μάλιστα προς όφελος του γεωργικού πληθυσμού, προς όφελος των καταναλωτών και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται και με αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε, αν ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα, πιστεύω ότι και η γνωμοδότησή μου θα είναι ισορροπημένη και περιεκτική. Αυτά λοιπόν και καλό τους και οδησηγητές και τους συναδέλφους αν δεν έχουν αντίρρηση και αν τους βολεύει να έχουν μια σύντομη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών ήδη αυτή την Πέμπτη γύρω στη μία. Θα τους στείλω και mail για να οργανώσω και το πρόγραμμά τους. Η πρότασή μου είναι να συνεδριάσουμε την Πέμπτη γύρω στη Μία με τους και ηγητές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους και πραγματικά χαίρομαι και περιμένω με ανυπομονησία όλο και πιο λεπτομεριακές προτάσεις. Ευχαριστώ. Μέχρι 9 Δεκεμβρίου θα πρέπει να κατατεθούν οι τροπολογίες. Σε 9 Δεκεμβρίου λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, μην το ξεχνάτε και η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου. Αλλά μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου έχετε διορία για να υποβάλλετε τροπολογίες. Περνάμε στο επόμενο σημείο, κατάσταση ε, και εξελίξεις ε, των ε, διαπραγματεύσεων και των τριμερών διαλόγων. Θα ήθελα να δώσω πέντε λεπτά στον κάθε αρμόδιο για να μας ενημερώσει χωρίς συζήτηση μετά γιατί ήδη έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να συνεδριάσουν και οι συντονιστέ. Αυτή είναι η πρότασή μου λοιπόν. Μόνο πέντε λεπτά για ενημέρωση για τι τρέχουσε διαπραγματεύσει στου τρει αρμοδίου συζητητέ. Μην ξεχνάτε και την έκθεση που σας ανέφερα χθε που γίνεται στον τρίτο όροφο, επευκαιρία του Παγκόσμιου Έτους των Εδαφών δεν θα ήταν πρέπον να, να απουσιάζουν τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας από τόσο σημαντική έκθεση. Ο κύριος Άγγινιο. Πρόεδρε, πάντα σέβομαι το χρόνο που διατίθεται για τι αγορεύσει. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω ω για ένα σημείο εδώ, να μου επιτρέψετε ένα λεπτό αφού λάβουν το λόγο οι συγγητές, Σας παρακαλώ. Σα ευχαριστώ μάλλον θα γίνει. Ο κύριος Χόισλινγκ πρώτα. Ενημερώστε μας παρακαλώ για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Κύριε Πρόεδρε, ούτε καν μου χρειάζονται τα πέντε λεπτά, δεν έχω πολλά να πω. Μία μόνο συνάντηση τριμερούς διαλόγου έχει διεξαχθεί με τη Λουξεμβουργική Προεδρία του Συμβουλίου. Νομίζω όμως ότι έχουμε προχωρήσει, δηλαδή εξετάσαμε την ημερήσια διάταξη την ημέρα εκείνη και καθιερώσαμε κάποιες βασικές αρχές για να γίνει ο τριμερής διάλογος. Συμφωνήσαμε για τους ελέγχους, ότι αυτοί πρέπει να απλοποιηθούν και να βελτιωθούν. Συμφωνήσαμε επίσης ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή εναρμόνιση, η οποία λείπει για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού και βέβαια εμείς θέλουμε μάλιστα νέο κανονισμό. Συζητήσαμε πρώτα για το πεδίο εφαρμογής και σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσαμε, μιλήσαμε για τις βασικές αρχές και εκεί προχωρήσαμε αρκετά. Μετά φτάσαμε σε μια κάπως αμφιλεγόμενη ε, υπόθεση που είναι οι μικτές επιχειρήσεις. Συζήτηση που έχει διεξαχθεί και εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Συμφωνήσαμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν μικτές εκμεταλλεύσεις και αυτό το θέλει άλλωστε και η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. Αλλά χρειάζεται να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Δηλαδή οι μονάδες παραγωγής πρέπει να είναι ξεκάθαρα διακεκριμένες στις μικτές επιχειρήσεις. Ήρθαμε και στο θέμα των ελέγχων όπου όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η έλεγχη προβλέπει ο ε, κανονισμός πρέπει να διατηρηθούν. Ταυτόχρονα γίνεται και άλλος τριμερής διάλογος για τον οριζόντιο κανονισμό. Πρέπει λοιπόν εκεί να φροντίσουμε να περιληφθεί μια παραπομπή ότι δηλαδή οι έλεγχοι ρυθμίζονται στα ε, περί παραγωγής, δηλαδή στον κανονισμό περί παραγωγής. Και τέλος συζητήσαμε στη συνάντηση εκείνη και τους κανόνες περί εισαγωγών. Εκεί θέλουμε να επιτύχουμε την συμμόρφωση, compliance, για τις εισαγωγές, που κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε να ισχύσει ως θεμέλιο, όμως για πολλές εισαγωγές χρειάζονται και κανόνες εξαρέσεων. Εκεί πρέπει να προβλέψει κάποια πρόταση η Κομισιόν για ορισμένες χώρες δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζονται οι κανονισμοί μας περί βιολογικής παραγωγής. Στις 9 του μηνός θα διεξαχθεί ο δεύτερος τριμήρης διάλογος και θα πρέπει μετά να μπορέσουμε να περάσουμε και στην επόμενη βέβαια προεδρία. Είμαι όμως διακατέχομαι από την πεποίθηση ότι θα το επιτύχουμε και ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα προχωρήσουμε, ε, με πολύ γρήγορο ρυθμό. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά τα ζωοτεχνικά θέματα, έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος, κάπως ιδιαίτερη κατάσταση. Για μια φορά το Κοινοβούλιο υιοθέτησε πριν το Συμβούλιο τη θέση του. Και στην σύνταξη των τροπολογιών το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Εν γέννη έχουμε ευθυγραμμιστεί πολιτικά με τους μεγάλους στόχους. Ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς, διατήρηση των, ε, από τις ράτσες που κινδυνεύουν και να διατηρήσουμε τις ιδιαιτερότητες των ειδών, κυρίως όσον αφορά τον τομέα των ύπων. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε εδώ και 15 μέρες περίπου. Αφορούσε την οργάνωση τομέα, τους κανόνες για την ε, διαχείριση ε, των γεωλογικών ε, γραμμών, έλεγχος επιδόσεων και γενετικών χαρακτηριστικών. Παρεκκλήσεις για τα σπάνια είδη, υβριδικά ζώα κλπ. Εκτελέσεις των διαφόρων προγραμμάτων. Αυτές 85 95% των σημείων έκλεισαν όσον αφορά τις τυχε παραμενουν παραμένουν 2-3 για τα σημεία. Το θέμα τη υποχρέωση ή μείωση των εγκρίσεων των προγραμμάτων επιλογή από τα διάφορα είδη. Σίγουρα θα τεθεί και θέμα επικουρικότητα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Αίτια άρνηση από το πρόγραμμα επιλογή, συμμετοχή στο πρόγραμμα επιλογή πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ μη κατακαιρμάτιση των καθαρέμων αν δεν υπάρχει στο συντονισμός και αν δεν γίνονται σεβαστές οι πτυχές ε, των διαφόρων προδιαγραφών και εμπόριο, πώς αδειοδοτείται το εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τελικά. Η μάχη για τους κανόνες για την καταξιδότηση πράξης και τις εκτελεστικές πράξεις είναι κάτι που θα συζητηθεί στον τελευταίο τριμερή διάλογο. Μεθαύριο θα γίνει άλλος διάλογος. Τρεις συνεδρία τεχνικού επίπεδου έγιναν ήδη επέτρεψαν να προχωρήσουμε επί των σημείων που προανέφερα, που παρέμεναν εκρεμεί στον πρώτο τριμερή διάλογο. Ο τριμερή διάλογο δεν πρέπει να επιτρέψει να προχωρήσουμε όσον αφορά το ενδοευρωπαϊκό ε, εμπόριο και τι αγωγέ του τρίτε χώρε για τον επίσημο έλεγχο και τον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να υπογραμμίσω ότι το κείμενο του Συμβουλίου είναι, ε, έχει καλή ποιότητα νομική και οι θέσει του Κοινοβουλίου ελήφθη σε σημαντικό ποσοστό υπόψη όσον αφορά επισήμου ελέγχου φαίνεται σημαντικό να εξασφαλίζεται η επίσημη όλογχη, έλεγχη συγγνώμη, και η ποιοτική έλεγχη, να επικρατεί διαφάνεια και να μην δημιουργείται υπερβολικό άχθος όσον αφορά ε, την επιλογή των ζώων ε, και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ε, συνεργάζονται μεταξύ τους διοικητικά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις παρεκκλήσεων. Ο τομέας γενικά δεν είναι τόσο όσο ο, αυτός των τροφίμων, των τροφίμων και θα πρέπει τελικά να τροποποιηθούν οι διατάξεις που πρόβλεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Συμβουλίου, σεβόμενοι το πνεύμα ε, των αρχικών κειμένων. Αυτά ήθελα να σας πω. Pani poseł Κυρία Μακιντάιρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ενημερώσω για την επιτευθύσα πρόοδο, για τους τριμερείς διαλόγους, για το νέο κανονισμό, ε, για τα διάφορα παράστα των φυτών. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης συζητητές. Έκαναν πολλή δουλειά και σημειώνεται πρόοδος. Πέντε τριμερείς διάλογοι έλαβαν χώρα μέχρι τώρα και έχουν προγραμματιστεί άλλοι δύο, 8 Δεκεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε λοιπόν να πετύχουμε συμφωνία δεύτερης ανάγνωσης πριν το τέλος του έτους. Υιοθέτησε τη θέση του το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2014. Το Συμβούλιο φώνησε επί της εντολής αυτού μόνο τέλος Ιουνίου φέτος. Και το τροποποιηθέν κείμενο από πλευρά Συμβουλίου συμπεριλαμβάνει πολλές αλλαγές σε σχέση με την πρώτη ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρκετές είναι σημαντικές και πολιτικά και θεσμικά. Οι πέντε τριμερείς διάλογοι που έλαβαν χώρα. Εκεί σε αυτούς εξετάσαμε το κεφάλαιο 1 που αφορά το πεδίο εφαρμογής ορισμούς το κεφάλαιο 2 το συζητήσαμε, αφορούσε για την καραντίνα όσον αφορά αυτά τα παράστητα. Κεφάλαιο 3 με, αρχικά αφορούσε κα, αφορά την Ένωση και τη θέση της όσον αφορά ε, τα παράσιτα που δεν, αφορούν, δεν ε, συνεπάγονται καραντίνα μετά ποιοτικού ελέγχους κεφάλαιο 4 και 5 για την καταχώρηση των επαγγελματικών επιχειρηματών και την ιχνηλασιμότητα. Στου τελευταίου δύο τριμερεί διαλόγου πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα άρθρα του κεφαλαίου 6, πιστοποίηση φυτών, φυτο, φυτικών προϊόντων και άλλα αντικείμενα, κεφάλαιο 7 και κεφάλαιο 8 και όλες τις αιτιολογικές σκέψεις, άρα έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Από τα βασικά θέματα. Ποια είναι τα βασικά θέματα, πώς να εντοπίσουμε τα παράστα που έχουν προτεραιότητα, πώς θα καταχωρηθούν τα παράστα, καθεστώς εισαγωγών και το θέμα των εφαρμοστικών πράξεων και εξουσιοδότησης πράξεων. Ένας τομέας που μας προβλημάτισε ιδιαίτερα ήταν ο αριθμός των ε, παρασίτων που έχουν προτεραιότητες. Ε, το Συμβούλιο υποστήριζε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι προτεραιότητες δεν πρέπει να ξεπερνούν αυτά το 10% του συνολικού καταλόγου. Η, τροπολογία μας 40 ήθελε να διαγραφεί αυτό το αυθαίρετο 10% και διαπραγματευθήκαμε πάνω σε αυτές τις γραμμές διότι το όριο του 10% θεωρούσε το Κοινοβούλιο ότι ήταν κάτι αδικαιολόγητο και αυθαίρετο. Οπότε προτιμούσαμε ο περιορισμός των προτεραιοτήτων να περνά μέσω της θεσπίσεως κριτηρίων που θα αναφέρονται στο παράρτημα 2. Το Συμβούλιο δέχτηκε τη διαγραφή του 10% του ορίου αυτού, του 10%, αλλά οι διαπραγματεύσεις για το παράρτημα 2 και τα συμπεριλαμβανόμενα κριτήρια δεν έχει λήξει ακόμα. Επίσης, κάναμε και κάποια δουλειά όσον αφορά τις εφαρμοστικές πράξεις και τις κατεξισοδότησης πράξεις. Είναι επίμαχο το ζήτημα αυτό. Μέχρι κάποιο βαθμό έχουμε συμφωνήσει. Όμως απομένουν πολλά προς διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Μας βοήθησε πολύ για τις εφαρμοστικές πράξεις και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και τον εμπειρογνώμονα θέλω να ευχαριστήσω για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, τους εμπειρογνώμονες. Μας βοήθησαν πολύ. απομένουν τομείς προσκάλυψη. Όμως τρέφουμε ελπίδες για συμφωνία πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Σας ευχαριστώ κύριε Σάγνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σουηδή βιολογική γεωργοί με παρακάλεσαν να μεταφέρω εδώ ότι αντιμετωπίζουν μέγα πρόβλημα με τον νέο κανονισμό περί βιολογικής γεωργίας. Ψυχρή χώρα και αυτοί ε, φυτεύουν τις σαλάτες τους σε ε, υπερυψωμένα φυτόρια με τρόπο που ικανοποιούν τους ε, ε, κανονισμού που ισχύουν στην πατρίδα του και του καταναλωτέ του, όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να του απαγορεύσει να το πράξουν, που σημαίνει δεν θα μπορούν να, ε, να ικανοποιήσουν τι απαιτήσει των καταναλωτών και τελικά θα κλείσουν τα φυτωρία του. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στον τριμερή διάλογο και ίσω ακόμη και σε αυτό το προχωρημένο στάδιο των διαπραγματεύσεων να πρέπει κάτι να γίνει για την προστασία των ε, παραγωγών αυτών. Σας ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμη αυτή η παρατήρηση. Θέλει κάποιος οπωσδήποτε να λάβει το λόγο. Ε, κύριε Αγγιλέρα, αν θέλετε, ένα λεπτό μόνο όμως. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Πολύ σημαντική η ενημέρωση που μας έκαναν οι συγκητές για τα τρία αυτά θέματα. Εμένα με ενδιαφέρει και με απασχολεί ιδιαίτερα η εξέλιξη των συζητήσεων για τη βιολογική γεωργία, αυτά που μας είπε ο κύριος Χόισλινγκ. Μακάρι να διεκπαιρεωθεί το θέμα το συντομότερο δυνατό και να έρθει σε αίσιο πέρας, γιατί αυτό περιμένουν η Ευρωπαίοι παραγωγή και δι η Ισπανή παραγωγή. Ε, νομίζω ότι δεδομένων των συμφωνιών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επήγει η διεκπαιρέωση του θέματος. Είμαστε σε καλό δρόμο, όπως είπε ο κ. Χόισλινγκ, αλλά μας μένει πολύς δρόμος ακόμη. Και τα άλλα δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά και χαίρομαι που διαπιστώνουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Yes, thank you, Just Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω και εγώ και να υπερθεματίσω σε αυτά που είπε ο κύριος Άγνιο για τη βιολογική γεωργία. Και φυσικά όταν είναι παγωμένο το έδαφος είναι αδύνατο να, να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε καλλιέργεια. Γι' αυτό και έχουμε τα περιψωμένα φυτόρια. Αφήστε μας αυτή τη δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς και την υγεία των ζώων, θα ήθελα να εξετάσουμε εκ του σύνεγγε αυτό το θέμα, γιατί η έκβαση των τριμερών διαλόγων ίσω επηρεάσει πολύ σοβαρά της ε, συμφωνίες διεθνούς εμπορίου. Και θα ήθελα να αποφύγουμε ε, κακή νομοθεσία όταν η στρατηγική μας μιλά για ευνομοθετή. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ αυθαίρετες οι προτάσεις που προκύπτουν ε, στον τριμερή διάλογο και ίσως βλάψουν σημαντικά τις αγωγές. Ο τελευταίος παρακαλώ. Ένα λεπτό κι εσείς, αλλά τελευταίος μιλητής για σήμερα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό χρειάζομαι ούτως ή άλλως, όχι παραπάνω. Εγώ λαμβάνω μέρος στις συζητήσεις του τριμερούς διαλόγου για το νέο κανονισμό για την υγεία των φυτών. Α μην ξεχνούμε ότι είμαστε Επιτροπή Γεωργίας και θα πρέπει ω τέτοια να προσπίσουμε τα συμφέροντα των γεωργών μας και να υπερασπίσουμε την παραγωγή μας. Είχαμε τους τελευταίους μήνες ε, ε, πολλού πολλούς επιβλαβείς οργανισμούς σε πολλές καλλιέργειες ε, με τεράστια θνησιμότητα, ιδιαίτερα στα ελαιόδεντρα εξαιτία της ξυλέλα, ξυλέλα φαστιδιώσα. Και οι παραγωγοί έχουν πληγεί θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν τα δικά του συμφέροντα και ω Επιτροπή Γεωργίας να υπερασπίσουμε τους γεωργού μας που ζητούν έλεγχο ώστε να μην επιτρέψουμε στου επιβλαβείς οργανισμούς να βλάψουν ή και να εξολοθρεύσουν την ευρωπαϊκή παραγωγή. Ευχαριστώ. Φυσικά θα επαναρχόμαστε συστηματικά στα θέματα αυτά και θα ζητούμε από τους εισηγητές μας τακτική ενημέρωση για την πορεία των τριμερών διαλόγων γιατί πραγματικά αυτά τα τρία θέματα είναι πολύ σημαντικά. Ε, σας υπενθυμίζω 12.30 ε, ε, τα εγγένεια στον τρίτο όρφο της έκθεσης ε, για τα εδάφη. Και μην ξεχνάτε ότι στις 3 έχουμε δημόσια ακρόαση για τη βελτίωση των φυτών. Θα περάσουμε τώρα στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ να παραμείνουν στην αίθουσα μόνο οι συντονιστές και όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται